Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ. Συνεχίζουμε με το πρόγραμμα της συνάντησης της Επιτροπής μας με τις ψηφοφορίες. Βλέπω ότι υπάρχει απαρτία και έχουμε και τους εισηγητές, μερικούς εισηγητές μαζί μας και μπορούμε να αρχίσουμε με την ετήσια έκθεση 2015 για τα, την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμηση της απάτης. Η κυρία Τζουφρίντα είναι η συγγήτρια και αρχίζουμε με τη συμβαστική 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13, τροπολογία 13, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 13. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε για τις 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 10. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε με ονομαστική το τελικό κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται η γνωμοδότηση. 28 υπέρ και μόνο 8 αποχές. Άρα να σας συγχαρούμε. Το... Η επόμενη ψηφοφορία Είναι η διαδικασία απαλλαγής. Καλύτερα όταν είναι υπογραμμισμένο το κείμενο με κίτρινο μαρκαδόρο. Λοιπόν, γνωμοδότηση για τη διαδικασία απαλλαγής για το 2015. Η κυρία Μιχαήλοβα είναι η συγγήτρη και αρχίζουμε με την συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα. 48 ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία. 48. 48. Ελέγχουμε την 48. Πέρας. Ε, λυπάμαι, αλλά το ΕΛΚ έχει έναν υπεράριθμο. Άρα πρέπει να ακυρωθεί η ψηφοφορία. Τι γίνεται. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία ηλεκτρονικά 48. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. και εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τώρα. The next European semester for... Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, Ετήσια Ανάπτυξη συντονισμός, ετήσιο συντονισμός. Ο κύριος Χέκμαν είναι εισηγητής και αρχίζουμε με τη συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Αν θέλετε να ελέγξουμε, ωραία. Ελέγχουμε την 6 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. If you count them, if you count them, they are less. Νομίζω ότι είναι κάτω από 12 τα μέλη του ΕΛΚ. Άρα δεν υπάρχει. Υπάρχει υπεράριθμος. It is Okay. It is... Απορρίπτεται. Η 6. 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εννέα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17, 17. Ελέγχουμε την 17, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. 18. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Την 20, ναι, την ανέφερα. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 34 υπέρ, κατά αποχές ας ελέγξουμε την 34 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική η οποία και άρχεται. And the vote Πέρας. Και εγκρίνεται. Η γνωμοδότηση με 31 ψήφους υπέρ. Σας ευχαριστώ πολύ. And now. And now we go for the draft motion for. Πρόταση ψηφίσματος ε, για την καθυστερημένη ε, εφαρμογή των λειτουργικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, Επενδύσεων ο κύριος Νοβακόφ είναι ο εισήγητης. Αρχίζουμε με τη συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6 υπέρ, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 68. Υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε την 68. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ, κατά υπάρχει και μία προφορική, με συγχωρείτε. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Φαίνεται πως όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την 84 με την προφορική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 86. Α, καταπίπτει. Άρα φτάνουμε στην 89. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Με την προφορική, την προσθήκη της προφορικής υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Άρα ψηφίζουμε την 11 με την προσθήκη της προφορικής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τελικό κείμενο. ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. 33, ε, με 33 ψήφους υπέρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν το προσχέδιο και σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.

Παρακαλώ καθίστε, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη και χαίρομαι ε, γιατί μπορώ να καλωσορίσω τον κύριο Λεμέτ. The Director Γενικός Διευθυντής της Περιφερειακής και ε, Πολιτικής Άστεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι ήδη τον έχετε γνωρίσει πολλοί από σας, αλλά τώρα έχετε τη δυνατότητα να τον ε, καλωσορίσετε και εδώ στη δική μας συνάντηση. Κύριε Λεμέτρ, σας ε, Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. Θα συνεργαστούμε τα επόμενα δυόμιση χρόνια μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα γενεά της πολιτικής μας αυτής, περιφερειακής και αστικής, μετά το 2020. Και φυσικά θα προβληθούν και προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου από την Κομισιόν και θα έχουμε πολλές ε, δυνατότητες να συναντηθούμε. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά για την εισήγησή σας και στη συνέχεια θα υποβληθούν ερωτήσεις και μετά θα αρχίσουμε τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Έχετε το λόγο. Κυρία Μιχαήλοβα, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας. Οι ευχές σας, προς περιλαμβάνουν θα έλεγα και κάποιους λόγους αν θέλετε προστασίας των δικών σας συμφερόντων σε εισαγωγικά. Τι εννοώ με αυτό. Ήταν, είναι η στιγμή πάρα πολύ καλή που θα συζητήσουμε. Τους προηγούμενους μήνες είχα κάποιες ευκαιρίες να συναντηθώ με ορισμένα από τα μέλη της Επιτροπής σας ιδιαίτερα τον Οκτώβριο με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Επιτροπή Πολιτισμού. Αλλά ο Ιανουάριος είναι η καλύτερη στιγμή για να σας παρουσιάσουμε τις φιλοδοξίες μας και το πρόγραμμα εργασίας μας και να ακούσουμε από σας το ποιες είναι οι επιθυμίες σας και τι θα θέλατε να δείτε να κάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο. Η πρόθεσή μου στην παρούσα φάση δεν είναι το να προχωρήσω σε, σε σχόλια και σε λεπτομέρειες. Να πω μόνο ότι το 2017 θα είναι πραγματικά διαφορετικό από τα προηγούμενα. Και μετά από τη συζήτηση που θα έχουμε ίσως να μπορέσουμε να το ε, σχολιάσουμε κάπως περισσότερο. Σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας μας λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια παρουσίαση η οποία θα διαιρείται σε τρία επιμέρους θέματα. Το πρώτο είναι η εφαρμογή, δηλαδή η παρούσα περίοδος. Το δεύτερο είναι νομοθετικά θέματα, τα οποία είναι ήδη υποσυζήτηση. Και το τρίτο θέμα είναι ε, στρατηγική για μετά το 2020, μελλοντικές δηλαδή προτάσεις. Για τα θέματα της εφαρμογής. Δεν είναι σαφές το που ε, θα επιθυμούσαμε να βρισκόμασταν σε αυτή τη φάση. Έχουν περάσει τρία χρόνια από το 14 σχεδόν, από την αρχή δηλαδή της περίοδου 14-20 και οι φιλοδοξίες μας ήταν υψηλότερες. Υπάρχουν θετικά νέα τα οποία ήρθαν στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες. Υπάρχει μια σαφής επιτάχυνση στους ρυθμούς επιλογής προγραμμάτων τους τελευταίους μήνες. Και νομίζω ότι σε μία περίπου εβδομάδα θα έχουμε μία πλήρη επιβεβαίωση αυτού του ισχυρισμού γιατί στο τέλος του Ιανουαρίου κάθε χώρα θα μας στείλει τους ανανεωμένους αριθμούς, τα ανανεωμένα στοιχεία για το ρυθμό επιλογής. Συγκρίνοντας με αυτά τα οποία είχαμε τον μήνα Οκτώβριο, μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί ιδιαίτερως, θα υπάρξει ένα άλμα στο ρυθμό. Πέραν τούτου όμως, ε, δεν υπάρχει εδώ ιδιαίτερος χώρος για ικανοποίηση. Θα συνεχίσουμε εμείς ε, να χρησιμοποιούμε κάθε δυνατότητα την οποία έχουμε μπροστά μας, έτσι ώστε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, να εξακολουθήσουμε φυσικά να πιέζουμε τα κράτη-μέλη και να συζητάμε μαζί τους τα εμπόδια τα οποία συναντούν στην, στον τομέα της εφαρμογής. Πάντως οι προσδοκίες μας είναι ότι το 2017 θα είναι μια χρονιά εξομάλυνσης του ρυθμού εφαρμογής και ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε ιδιαιτέρως θα έλεγα, θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να συζητάμε τα θέματα του μέλλοντος από μια σχετικά καλή θέση. Νομίζω ότι στο τέλος του 2017 η εικόνα θα είναι σαφώς βελτιωμένη συγκρίνοντας με το τέλος του 2016. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα θέσω σήμερα είναι τα τρέχοντα νομοθετικά θέματα, οι νομοθετικοί φάκελοι που είναι υπό εξέταση. Υπάρχουν δύο που γνωρίζετε πολύ καλά. Ο πρώτος είναι η πρόταση πακέτο Omnibus, προφανώς μια περίπλοκη και ιδιαίτερος τεχνική πρόταση, η οποία όμως νομίζω ότι με κάποιες ε, θα έλεγα προσπάθειες ε, να ξεκαθαρίσουμε τους στόχους ε, θα είναι πολύ χρήσιμη. Πρώτος στόχος, κατά τη διάρκεια της παρούσης περίοδου, να πετύχουμε κάποιο ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απλοποίησης για τους δικαιούχους. Νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Νομίζω ότι κάναμε αρκετά βήματα προς τα εμπρός χωρίς να διαταράξουμε τα συστήματα τα οποία είχαν τεθεί σε λειτουργία. Είχαμε εμπνευστεί από τις προτάσεις της ομάδας υψηλής εργασίας για την απο, απλοποίηση της οποίας προεδρεύει ο κύριος Κάλλας. Ε, νομίζουμε ότι τελικά τα τελικά στοιχεία της πρότασής μας θα γίνουν δεκτά από τους συνομοθέτες και το λέγω αυτό γιατί σήμερα δεν είμαι απόλυτα βέβαιος, ιδιαίτερα βλέποντας ποια είναι η δυναμική στο εσωτερικό του Συμβουλίου, υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις θα έλεγα, τις οποίες ομολογώ ότι δύσκολα μπορεί να κατανοήσει κανείς, αλλά παρόλα αυτά πέραν αυτού μάλλον και με το Συμβούλιο και με εσάς εδώ Είμαστε απολύτως διαθέσιμοι για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις σχετικά με την ύπαρξη μιας πραγματικά περίπλοκης πρότασης έτσι ώστε να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση το θέμα της επίτευξης ενός θετικού αποτελέσματος είναι κυρίως και θέμα θα έλεγα χρονισμού. Η δουλειά μας έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατόν να έχουμε την δυνατότητα να δουλέψουμε πάνω σε ένα συναποφασισμένο ε, κείμενο ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Χτες έγινε μια πολύ καλή συνάντηση ανάμεσα στην κυρία Κρέλα και τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο ε, και πέραν αυτής της συνάντησης πάντα είμαστε πλήρως διαθέσιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης ε, σε μια πιο πρόσφατη πρότασή μας η οποία αν θέλετε ήρθε στην επικαιρότητα από τα τελευταία γεγονότα, δυστυχώς πολύ αρνητικά γεγονότα, τραγικά γεγονότα. Αναφέρομαι στην πρόταση τροπολογίας που θα επιτρέψει στην πολιτική συνοχή να επιδεικνύει και μεγαλύτερη αλληλεγγύη σε περιπτώσεις όπου έχουν υπάρξει σοβαρότατες φυσικές καταστροφές εμείς εμένουμε στην Ρέγγιο ότι έχει φτάσει πλέον η στιγμή να δείξουμε την αλληλεγγύη μας με ουσιαστικό τρόπο και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και ταχύτατα. Συνεπώς λοιπόν ελπίζω ότι λόγω ακριβώς και του απλού χαρακτήρα της πρότασης μπορούμε να στοχεύουμε για ένα ταχύτερο χρονοδιάγραμμα από ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί στα, στο παρελθόν. Και τέλος, ο τελευταίος τομέας τον οποίο θα θίξω είναι η δουλειά μας για το μέλλον. Με μεγάλη ικανοποίηση, όχι μόνο σήμερα, αλλά και εδώ και λίγες εβδομάδες, ενημερώθηκα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να υιοθετήσει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και ότι η έκθεση αυτή, αυτό θα φανταζόμουν εγώ σαν κάτι το ιδανικό, θα κυκλοφορήσει πριν από την σημαντική στιγμή το 17 για την πολιτική συνοχή το Φόρουμ Συνοχής, το οποίο θα οργανωθεί στα τέλος του μηνός Ιουνίου. Θα ήταν λοιπόν ευκταίο η δική σας έκθεση πρωτοβουλίας, η οποία θα αποτελέσει ένα από τα σημεία αναφοράς αν θέλετε, της διοργάνωσης αυτής του φόρουμ να είναι διαθέσιμο νωρίτερα και είμαι πολύ ικανοποιημένος και για το ότι οργανώσατε πάνω σε αυτό ήδη σήμερα το πρωί ένα workshop, ένα εργαστήριο επεξεργασίας θέσεων. Εμείς από τη δική μας την πλευρά βέβαια αυτό το οποίο θέλουμε είναι να προπαρασκευαστούμε σωστά για να καταθέσουμε τις μελλοντικές προτάσεις. Και αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι να έχουμε την δυνατότητα να διαθέσουμε τις προτάσεις μας σε αρκετά σημαντικούς τομείς για το μέλλον. Ε, θα αναφερθώ στους τομείς αυτούς ε, με χρονολογικό τρόπο, όπως ακριβώς θα τους παρουσιάσουμε. Το πρώτο έγγραφο πρόταση που θα δείτε από μας αφορά την εξάντε ερεσιμότητα, την εκ των προτέρων ερεσιμότητα. Το έγγραφο αυτό θα κυκλοφορήσει στο τέλος του μηνός Μαρτίου. Βασικός στόχος του εγγράφου αυτού είναι όχι να κάνει μια πλήρως τελική αποφασιστική αξιολόγηση ε, του τι έχει, ε, ε, θα έλεγα, παράξει αυτός ο νέος μηχανισμός, αλλά ένα, εν πάση περιπτώσει, έλεγχο και να δούμε ποια είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο ισχυρισμός μας λέγει ότι η αξιολόγηση αυτή θα είναι θετική. Όπως είπα δεν θα είναι η τελική αξιολόγηση, διότι είναι σαφές ότι κάποιες αιρεσιμότητες σε εισαγωγικά εξάντε δεν θα έχουν εκπληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου. Αλλά δεν είναι αυτό το σημείο που θα μας απασχολήσει, ελπίζω. Αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι το σύνολο των μεταρρυθμίσεων, διότι περί αυτού πρόκειται, ε, το σύνολο των διοικητικών ε, διακανονιστικών ρυθμίσεων τις οποίες θα αναλάβουν να φέρουν εις πέρα στα κράτη-μέλη και μάλιστα σε ένα σύντομο χρονικό σχετικά διάστημα έτσι ώστε από τη μία να διασφαλίσουμε ότι οι δαπάνες στον τομέα της συνοχής θα είναι υψηλότερας ποιότητας από ό,τι στο παρέλθον και από την άλλη να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ε, σε περισσότερες μεταρρυθμίσεις οι οποίες να διαμορφώνουν ένα περιβάλλον φιλοαναπτυξιακό θα θέλαμε λοιπόν εμείς να το εξετάσουμε αυτό το θέμα σύντομα, γιατί ξέρετε είναι ιδιαίτερο σκενοφανές αυτό που γίνεται. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε εμείς για πρώτη φορά. Αλλά αν εξετάσει κανείς τα γενικώς διαθέσιμα μέσα δημοσιονομικής φύσεως, δεν θα δει έναν αντίστοιχο τέτοιου τύπου μηχανισμό. Και αν εξετάσει κανείς το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τον τρόπο λειτουργίας του ε, Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, οι συστάσεις αναχώρα, οι εξειδικευμένες αναχώρα συστάσεις, δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε μορφή κινήτρων, αν θέλετε, εκτός από αυτά τα οποία ήδη συμπεριλαμβάνονται στην πολιτική συνοχής, της ρεσιμότητες εξάντε, όπως επίσης και μία πρώτη σειρά μέτρων μακροαιρεσιμότητας. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε σε μια σωστή αξιολόγηση γιατί η διάρθρωση των μεταρρυθμίσεων στο μέλλον είναι κάτι το ιδιαίτερο κρίσιμο. Και ο τρόπος με τον οποίο στο μέλλον εμείς θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στον τομέα των μεταρρυθμίσεων αυτών και να διαμορφώσουμε στη συνέχεια τις νέες πολιτικές είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει τον πυρήνα των συζητήσεών μας. Αυτό ήταν το πρώτο έγγραφο. Το δεύτερο έγγραφο θα κυκλοφορήσει και αυτό στο τέλος του μηνός Μαρτίου. Το έγγραφο αυτό αναφέρεται ε, στην λεγόμενη πρωτοβουλία για τις περιοχές που παρουσιάζουν χρονική ιστέρηση. Έχουμε εξετάσει δύο ε, τύπους περιφερειών που παρουσιάζουν κάποιες τέτοιες υστερήσεις, αν θέλετε. Οι πρώτες είναι οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε εδώ στοχεύσει δύο περιοχές στην Πολωνία και δύο στην Ρουμανία. Ε, η δεύτερη μορφή περιφερειών που μας ενδιαφέρουν είναι αυτές οι οποίες πραγματικά αρνούνται να συγκλίνουν. Ε, εδώ το θέμα δεν είναι υποχρεωτικά οι χαμηλότεροι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης που έτσι κι αλλιώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα έλεγα επί δεκαετίες προσπαθούμε να παρατηρήσουμε και να ορίσουμε. Αυτών των δύο ειδών οι περιοχές λοιπόν έχουν όπως είπα διαφορετικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζουν διαφορετικές προκλήσεις Και αυτό θα προσπαθήσουμε με το έγγραφο αυτό που θα κυκλοφορήσουμε να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι μετά από όλες τις έρευνες και τις αναλύσεις που έχουμε κάνει θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε την πολιτική μας αποτελεσματικότερη. Ιδιαίτερα για αυτές τις περιφέρειες οι οποίες επαναλαμβάνω ότι μέχρι σήμερα και παρά τις σημαντικότατες χρηματοδοτικές ενισχύσεις επί δεκαετίες θα έλεγα δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν και δεν έχουν καταφέρει να γυτνιάσουν του επίπεδου των υπολείπων περιφερειών. Η τρίτη ανακοίνωση είναι η λεγόμενη ευφυής εξειδίκευση, στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευση, το μήνα Μάιο. Όλα αυτά τα οποία σας λέγω θα γίνουν και θα ολοκληρωθούν πριν από το φόρουμ για την ε, ε, συνοχή. Νομίζω ότι και αυτή η ανακοίνωση όπως και η αντίστοιχη για τις εξάντερες ημότητες θα μπορέσουν να μας ε, δώσουν την εικόνα του πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις ευφυείς αυτές στρατηγικές, σε ποιους τομείς στρατηγικής φύσεως θα πρέπει να σταθούμε και τέλος <clears throat> πώς θα συμπληρώσουμε τα μέτρα αυτά έτσι ώστε να μπορέσουν να παράγουν το είδος των αποτελεσμάτων τα οποία εμείς θεωρούμε ευκταία. Ε, σαν παράδειγμα η διάσταση της συνεργασίας ανάμεσα στις στρατηγικές εφιούς εξειδίκευσης που δεν έχουν αναπτυχθεί με συστηματικό τρόπο σε όλες τις χώρες. <clears throat> Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Έχουμε προχωρήσει στον σχεδιασμό ορισμένων θεματολογικών πόλων, οι λεγόμενες θεματολογικές πλατφόρμες πάνω στις οποίες θα χτίσουμε. <clears throat> Υπάρχει και το φόρουμ φυσικά, το ίδιο το φόρουμ δεν είναι ένα απλό έγγραφο, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη συνοχή κατά τη διάρκεια του έτους και περιμένουμε ότι οι συζητήσεις για το μέλλον θα γίνουν πιο ενδιαφέρουσες και αποφασιστικές. Από την άλλη πλευρά, μετά το καλοκαίρι δηλαδή, ε, θα βγάλουμε μία ανακοίνωση για τα διαμεθοριακά εμπόδια. Αυτή η ανακοίνωση θα εξετάζει το θέμα των εμποδίων αυτών ε, με τον ευρύτερο δυνατό φακό, κάθε φύσεως δηλαδή εμπόδια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα περιοριστεί πλήρως στα παραδοσιακά μέτρα αξιολόγησης της ε, συνοχής, αλλά θα είναι μια προσπάθεια έβρεσης κάθε τρόπου και εντοπισμού κάθε τρόπου έτσι ώστε να ε, μπορέσουμε τις τροχοπέδες αυτές στην πρόοδο των πολιτών να τις απομακρύνουμε. Θα υπάρξουν δύο περαιτέρω ανακοινώσεις. Καταρχάς, η στρατηγική για τις απότερες περιφέρειες είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπιστεί επίσης. Πιστεύουμε ότι η στρατηγική αυτή για τις απομεμακρυσμένες περιοχές, οι απότερες περιοχές θα δημοσιευθεί τον μήνα Οκτώβριο. Και στο τέλος του 2017 ξέρετε ότι περιμένουμε και την τελική έκθεση για τη συνοχή. Είναι μια έκθεση την οποία απαιτεί η συνθήκη να παράγουμε ανατριετία. Πιστεύουμε ότι είμαστε αρκετά ικανοί στην παρούσα φάση να παράγουμε την έκθεση αυτή και ε, εφόσον μας το επιτρέψουν οι συνθήκες σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση αυτή για να ξεκαθαρίσουμε λίγο την ρητορική μας σε σχέση με το τι περιμένουμε να γίνει μετά το 2020. Τελειώνοντας, θα σταθώ στο θέμα της επικοινωνίας. Εγώ είπα ότι το 2017 είναι μια χρονιά διαφορετική από το παρελθόν και ότι το 2017 θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και στον τομέα της επικοινωνίας, επικοινωνίας της Ευρώπης γενικά και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας της πολιτικής συνοχής. Και αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε από κοινού με τους υπόλοιπους θεσμικούς εταίρους, με τα μέλη φυσικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών και με τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές. Αυτά. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πληρέστατη αυτή παρουσίαση. Σας ακούσουμε τώρα ερωτήσεις και σχόλια των συντονιστών από τις πολιτικές ομάδες, ο κύριος Φανίστελ Ρούι. Ευχαριστώ πολύ. Νέα χρονιά, νέα ομάδα, πολλά υποσχόμενοι πρέπει να πω, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Πολύ σημαντικό αυτό για την ανακοίνωσή μας. Μας δίνει τροφή σκέψης και αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε. Ξέρω ότι θα μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι, οπότε θα είμαστε σύντομο. Δύο παρατηρήσεις λοιπόν για την ε, ορατότητα, σε αυτό που καταλήξατε δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω μάθει, είναι ως συλλογικό όργανο μία και ενιαία. Και μοναδική. Όχι επαγωριστών βέβαια. Αυτό που βλέπω πάντως από τη στρατηγική την επικοινωνιακή είναι για μένα μεγάλες διαφορές. Βλέπουμε ότι η εικόνα είναι τελείως διαφορετική, δεν την υιοθετεί ο πολίτης πλέον ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Είναι σαν να είμαστε σε ένα σταθερό ποδήλατο, στατικό ποδήλατο και να λέμε μια χαρά τα πάω, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να ανέβουμε και την ε, πλαγιά, την ανηφόρα. Δεν ξέρω αν η εικόνα με το ποδήλατο σας εμπνέει. Πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να ανέβουμε την ε, πλαγιά και πάνω απ' όλα πρέπει να πάμε και πιο γρήγορα. ενώ οι άλλοι έχουν καβαλήσει πύραυλο και πετάνε. Άρα λοιπόν και το θέμα της επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα και αν έχουμε καλές ιδέες από το κοινόβουλο, θα είναι σκόπιμο να τις ε, κοινοποιούμε, βεβαίως ε, με τα νομικά όρια που προβλέπονται, αλλά πρέπει να μπαίνουν και στο όμνιμπους χωρίς να το διαταράσουν. Και νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Γιατί μάλλον κοιτάμε το έδαφος που βρίσκεται από κάτω μας αντί να κοιτάμε μπροστά εκεί που πρέπει να πάμε. Και κάτι ακόμα. Πρέπει να μας απασχολήσει το εξή. Θα δεχθώ βεβαίως την πρότασή σας για την αλληλεγγύη, σεισμοί στην Ιταλία και όλα αυτά που αναφέρατε. Βεβαίως. Το έχουμε συστήσει και στην Ολομέλη, έχουμε κάνει ψήφισμα, ήρθε η κυρία Κρέτσου, τα είπαμε όλα. Η εντύπωση όμως που είχα εγώ, για να είμαι ειλικρινή, ήταν ότι οι ειδικέ περιστάσεις σημαίνουν και ειδική αντιμετώπιση. Πολύ καλά. έτσι και 100% να δοθούν στην Ιταλία. Ξέρουμε βέβαια ποια είναι η κατάσταση τώρα, δεν ξέρουμε που θα φτάσουν σε κανένα δύο μήνες, έτσι. Είναι ιδιαίτερη η κατάσταση λοιπόν. Αλλά τώρα βλέπω μια πρόταση τη επιτροπή που με έκανε να αναπηδήσω. Γιατί δεν πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίσταση. Βλέπω να ανοίγουν τα κριτήρια της αλληλεγγύης προς τα πάντα. Και τους πάντες. Και οι κάτω χώρες, αν έχουν κάποια τέτοια περίσταση. Αλλά εμείς δεν το χρειαζόμαστε. Αλληλεγγύη, η αλληλεγγύη θα πρέπει να γίνεται κατόπιν ετήσεως και με βάση τις ανάγκες του καθενός. Κουστούμι δηλαδή. Και αν σας ρωτήσω, μπορείτε να αποσύρετε αυτές τις προτάσεις και να έρθετε με μια πρόταση αλληλεγγύης ειδικά για την Ιταλία, θα το δεχθώ. Αλλά αυτό που κάνετε τώρα, 100% άνοιγμα της αλληλεγγύης, διαταράσσει την πολιτική μας και δεν είναι και σύμφωνα με τις αρχές μας. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλω να σας μεταφέρω και ευχαριστώ. Κύριε Κρέου. Κρέλ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική Διευθυντά αναφερθήκατε στη διαδικασία Omnibus. Φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε να μείνετε λίγο περισσότερο στην Επιτροπή μας όταν μετά από τη δική σας παρέμβαση θα συστήσουμε για πρώτη φορά την πρότασή μου το, την αντίληψή μου για ένα σχέδιο εκθέσεως ε, που θα συστήσουμε για πρώτη φορά. Εάν όμως ε, δεν μπορείτε να κάτσετε παραπάνω, τότε να σας δώσω το έγγραφο. Η Επιτροπή έχει στην πολιτική της συνοχής βάλει ένα-δύο πραγματάκια, έχει συμπληρώσει. Γιατί αν ήταν μια ολοκληρωμένη πρόταση, θα το δεχόμαστε βεβαίω στο κοινοβούλιο εδώ. Μιλάτε όμω για περιπτωσιολογία και με αυτήν πάτε να κάνετε ε, γενικευμένε αλλαγέ στην πολιτική. Έχω αμφιβολίε σε κάποια σημεία βεβαίω. Δεν ξέρω αν θα με ακολουθήσουν κάποιοι συνάδελφοι στις προτάσει που θα διατυπώσω, αλλά η διαπραγμάτευση με αυτά που μα λέτε δεν διευκολύνεται η κυρία Γκρέσλε έχει προτείνει ένα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα τα καταφέρουμε. Και γνωρίζω ότι τα κράτη-μέλη έχουν και από πλευρά τους ε, επιφυλάξει και εμβολίες. Δεν ξέρω αν θα τόσο απλά τα πράγματα για σας. Και δεν ξέρω αν ε, η Επιτροπή διευκολύνει το έργο της ε, βάζοντας τόσο διαφορετικά πράγματα, ειδικέ προτάσεις και ταυτόχρονα ε, ολικές αλλαγές της πολιτικής στην ίδια πρόταση. Επικαλεστήκατε την αλληλεγγύη, αυτό που ανέφερε και ο Λάμπερτ ε, για την περίπτωση φυσικών καταστροφών. 26 σχεδόν χρόνια είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εγώ Προερχομένη από την Ανατολική Γερμανία πρέπει να πω ότι πάντοτε ερχόμουν ε, με έκπληξη να αντιμετωπίσω τις προτάσεις για την πολιτική της συνοχής και το αίτημα για την ελληνική. Γιατί τότε πάμε για 100% συγχρηματοδότηση, μάλλον χρηματοδότηση, Οπότε έχουμε να κάνουμε με ανέγερση γέφυρας χωρίς να βρίσκεται ποτάμι από κάτω ή με ανέγερση μιας ε, γέφυρα και άλλες τέτοιες ανοησίες που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Και φαίνεται ότι αυτό βλέπουμε να συνεχίζεται, να συμβαίνει αυτή η μπαλαβή Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι λοιπόν, δεν πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Θέλουμε μια υγεία συγχρηματοδότηση, όσο δύσκολη και είναι αυτή. Ε, και βεβαίω όταν υπάρχουν εξαιρετικέ και έκτακτες περιπτώσεις θα γίνονται πιο ήπια τα μέτρα και οι προϋποθέσεις. Αλλά όταν για κάθε φυσική καταστροφή προτείνεται να ε, εξασφαλιστεί η δυνατότητα για παρέκβαση από κάθε αρχή της, αρχής της, της πολιτικής της συνοχής, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας χωρίς να χρειαστεί να βάλει το χέρι στην τσέπη θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν νομίζω ότι βοηθάει μια τέτοια πρόταση. Και η πρόταση του Λάμπερτ, ε, Φανίστριλ Ρόι, να αποσύρεται αυτή σας την πρόταση, είναι για μένα πολύ επικοδομητική. Καμία σχέση δεν έχει αυτό με το αν θέλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη ή όχι. Αν επικρατεί δηλαδή το πνεύμα τη αλληλεγγύη. Αντιθέτω, πιστεύω ότι υπάρχουν ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν με διαφορετικού τρόπου και βεβαίω για την αλληλεγγύη όποιο θέλει να την επιδείξει νομίζω ότι θα αναγνωρίσει πω εμεί εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακή πολιτική. είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Άλλωστε αυτό είναι και η πολιτική τη συνοχή, αυτό είναι το νόημά τη, Να δείξουμε αλληλεγγύη στι περιφέρειε. Επίσης, περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω τι συγκεκριμένο νόημα θα έχει αυτή η πρωτοβουλία για το lagging behind. Καθυστέρηση. Τι σημαίνει μια περιφέρεια δεν θέλει, λέτε, να αναπτυχθεί στην πραγματικότητα ή μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν είσαι θέση να αναπτυχθεί περαιτέρω. Ένα παράδειγμα. πολύ συχνά ακούμε να λένε «Αχ, στη Σικελία να δώσουμε επιδοτήσεις, ενισχύσεις, αφού δεν τις θέλουν, ε, δεν θέλουν την ανάπτυξη». Να μην δίνονται λοιπόν ενισχύσεις στη Σικελία και τότε τι θα κάναμε σε αυτήν την περίπτωση. Μια περιοχή όπως η Σικελία, μόνο ενδεικτικά την αναφέρω, δεν θα έχει μειώσει τη διαφορά της σε σχέση με άλλες περιοχές. Άρα τι είναι τι θέλουμε να πούμε και τι ε, μήνυμα αποστέλουμε όταν λέμε «Α, η τάδε περιφέρεια ή η η δυναμη περιφέρεια δεν θέλει να αναπτυχθεί περαιτέρω». Ελπίζω να σας έχω παρερμηνεύσει. Γιατί είναι δυνατόν να βάλουμε στον άλλον σφραγίδα «Εσύ δεν θέλεις να προχωρήσεις». Σε εποχές ευρωσκεπτικισμού καλπάζοντος δεν βοηθάνε τέτοιες δηλώσεις. Το Νοέμβριο με χαρά είδαμε τις πρώτες γραπτές προτάσεις για τη μελλοντική πολιτική της συνοχής. Ακριβώς την κατάλληλη στιγμή μάλιστα κατατίθενται. γιατί πρέπει πια να ξεκινήσουμε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο και με τα χρονοδιαγράμματα όπως προβλέπονται για τα επόμενα χρόνια τα όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως προκλήσεις και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό και το Brexit και επίσης το 2019 πάλι ευρωεκλογές, ε, νέα επιτροπή στη συνέχεια το 2020 και θέλουμε ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε τη μελλοντική πολιτική της συνοχής. Κάθε μήνα βλέπουμε να έρχονται νέες πληροφορίες. Νομίζω ήταν καλό να ενημερωνόμαστε πιο έγκαιρα. Είναι πολύ καλή η έκθεση τη συναδέλφου για τη μελλοντική πολιτική της συνοχής, εκφράζει τις δικές μας θέσεις και ελπίζω να δείξετε και εσείς διάθεση έγκαιρη συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και έτσι η Επιτροπή να αφουγκραστεί κάποιες από τις συστάσεις και τις συμβουλές του Κοινοβουλίου. Να δούμε μια καλύτερη συνεργασία στην προπαρασκευή των νομοθετικών προτάσεων. Γι' αυτό άλλωστε ξεκινήσαμε με την έκθεση πρωτοβουλία. Τη βάλαμε στο χρονοδιαγραμμά μα και ελπίζουμε ότι θα έχουμε στα τέλη Ιουνίου μια διεξοδική συζήτηση για το Ταμείο Συνοχή. Για πρώτη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Από τους στηρητικούς μεταρρυθμιστές δεν βλέπω. Ο κύριος από την ε, ομάδα των φιλελευθέρων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεστε εδώ για να έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποια ε, επιπρόσθετα σχόλια στην εισήγησή σας. Πιστεύω να μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε τις, ε, το πλαίσιο αυτό των κοινών διατάξεων και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για φυσικές καταστροφές σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να έχουμε μία Στη διαδικασία, μια επίγουσα διαδικασία αντιμετώπισης, γιατί αυτή είναι και η πρόθεση του νομοθέτη. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Αυτή είναι και η πρώτη μου αντίδραση ως προς τα λόγια σας για γρήγορη έγκριση. Βεβαίως θα τηρηθούν όλοι οι δημοκρατικοί κανόνες. Δύο ερωτήσεις. Σήμερα μιλήσαμε για τα χρηματοοικονομικά μέσα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρθηκε σε αυτά. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ε, για το 2017, ποιες είναι οι δεσμεύσεις, υπάρχει κίνδυνος και πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε εσείς το θέμα αυτό του decommitment. Νομίζω ότι το συζητήσαμε αυτό, συνέργειες, απλοποίηση και το θέμα γενικότερα της απαλλαγής από υποχρεώσεις. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ε, οι γενικές διευθύνσεις να μπορέσουν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι θα γίνει λοιπόν με το περιεχόμενο αυτής της σύμβασης, θα αποσταλεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάνα, ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον ε, Γενικό Διευθυντή που παρευρέθηκε στην ε, συνεδρίασή μας και γιατί μας δίνει την ε, δυνατότητα να γίνει αυτή η συζήτηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο κανονισμός Omnibus ε, μαζί με την ε, πολιτική συνοχής. Και θα ήθελα να αναφερθώ στην Κωνσταντσε Κρέλ, δηλαδή στις επικρίσεις της ως προς την ε, Επιτροπή για τον κανονισμό Omnibus. Νομίζω ότι ο κανονισμός αυτός, ο Omnibus, είναι ιδιαίτερα περίπλοκος. Οι προκλήσεις είναι πολλές και επειδή πιέζει ο χρόνος, αυτό δεν μας βοηθά για να γίνει μια σωστή συζήτηση. Και βέβαια μέσα στους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού. Γι' αυτό λοιπόν εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, η ουσία, το περιεχόμενο του κανονισμού Omnibus, η δυνατότητα πάνω απ' όλα της απορρόφησης ε, χωρίς περιορισμούς ε, των κονδυλίων της συνοχής. Και θα ήθελα πολύ συγκεκριμένα να σας ρωτήσω στην προσεχή περίοδο, μετά το 2020 δηλαδή. Η, τα μεγάλα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής πώς μπορείτε να το διασφαλίσετε. Η αρχή της εταιρικότητας, η εταιρική σχέση παραδείγματι με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο σχεδιασμό και την οργάνωση της πολιτικής της συνοχής, ε, στόχευση, Στόχη Ευρώπη 2020, πώς θα τους εξυπηρετήσει η πολιτική συνοχής. Αλλά και θέματα που είδαμε στη σημερινή μας, στην πρωινή μας ε, ε, συνεδρία στο εργαστήριο αυτό που κάναμε ε, τα ποσοστά της ενίσχυσης που μπορούν να δεσμευθούν φερειπίν για, για τον κοινωνικό αποκλεισμό, για, την, για τα αστικά κέντρα, για την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά δεν τα βλέπουμε στις προτάσεις σας. Και ιδιαίτερα για την προστασία από τις κλιματικές αλλαγές, οπωσδήποτε χρειάζονται βελτιώσεις εδώ στη στόχευση πώς μπορούν, όπως είπα, να διασφαλιστούν οι, τα επιτεύγματά μας μέχρι τώρα. Η κυρία Κρέλλα και άλλοι ανέφεραν ότι χρειάζεται ενισχυμένη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώς στο θέμα των διαοργανικών διαπραγματεύσεων. Να οργανωθούν, παραδείγμα, τη σημεία επαφής, ε, ε, σύνδεσμοι επικοινωνίας, και άλλη μία ερώτηση, τελευταία και ίσως άσχετη, αλλά πολύ σημαντική ως προς την ουσία για τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια σας απασχολεί ένα ενδιαφέρον θέμα. ΑΕΠ και πέραν αυτού, GDP and beyond. Ε, νέοι δηλαδή δείκτες που φαίνεται να είναι διατεθειμένη να εισαγάγει και να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μέτρηση ιδιαίτερα των αποτελεσμάτων της περιφερειακής πολιτικής. Εγώ δεν ήθελα να δω τι στοχεύετε, τι σκοπεύετε να κάνετε. Όχι μόνο το ΑΕΠ λοιπόν, αλλά και ενδεχομένως άλλοι δείκτε. κριτήρια επιμερισμού, ισότητας, ε, κοινωνικής δικαιοσύνης θα ενσωματωθούν στους δείκτες γιατί υπήρξαν στο παρελθόν, στα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερω ενδιαφέρουσε προσέγγιση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν πιο πολλέ πληροφορίε για το GDP and Beyond. Και αν μου επιτρέπετε, μια σύσταση ή επιθυμία, μια ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τη Γενική σα Διεύθυνση. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για τη δουλειά μα. Η Πρόεδρο. Ευχαριστώ, κυρία Ντεμάτο. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ είστε ακριβώς ενήμεροι. Θα αναφερθώ και εγώ στη μεγάλη τραγωδία του σεισμού που φαίνεται να ε, συγκλονίζει τους συναδέλφους που έλεγαν το λόγο πριν από μένα. Βεβαίω και είναι ευπρόσδεκτη πρόταση τροποποίηση του κανονισμού από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για το περιστατικά της 30ης Νοεμβρίου. Ιδιαίτερα αναφέρεται για το σεισμό η αναθεώρηση του κανονισμού για την περίοδο 2014-2020 και η πρόταση για εισαγωγή της δυνατότητας πλήρους χρηματοδότησης, 100% χρηματοδότησης, της ανοικοδόμησης και της αποκατάστασης περιλαμβανομένης του της πολιτιστικής κληρονομιάς. Βέβαια στο δημοσιονομικό, στο τεχνικό δελτίο αναφέρεται ότι θα πρέπει να έχει ουδέτερο προς τον προϋπολογισμό επίπτωση αυτή η πρόταση. Δεν θα πρέπει δηλαδή να επηρεαστεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης. Λοιπόν, βεβαίω και υποστηρίζουμε την πρόταση, είμαι ικανοποιημένη και μάλιστα θα επαυξήσω γιατί το Δεκέμβριο του 2016 το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα για το σεισμό και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει αίτη περαιτέρω και δεδομένη τη πολύ σοβαρή κατάστασης ζητεί από την Επιτροπή να αποκλείσει από τον υπολογισμό του εθνικού ελλείμματο τη Ιταλίας σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητα και ανάπτυξη τα δαπάνε ε, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αυτών ε, ε, περιστάσεων, αλλά και την αποκατάσταση και σταθεροποίηση. Άρα και σε αυτό το θέμα και στην πρόληψη και αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων. Μπορείτε να μα πείτε ποια είναι ποιος είναι ο γενικό προσανατολισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα συγκεκριμένα αυτά σημεία και πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να λάβει υπόψη τι θέσει που τον προηγούμενο Δεκέμβριο εξέφρασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Έξι ακόμη συνάδελφοι, ναι. Στον κατάλογο, επτά. Ναι, εσείς πρώτος, εσείς πρώτος. Θέλετε τώρα να απαντήσετε εσείς, κύριε Λεμέτρο, και να ακούσουμε μετά τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ωραία. Σας δίνουμε το λόγο για να απαντήσετε και θα συνεχίσουμε με τον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στα διάφορα ζητήματα που έθιξαν οι ευρωβουλευτές με τη σειρά τους. Αλλά ίσως οι απαντήσεις μου να ισχύουν ε, για διάφορα σχόλια που έγιναν, δηλαδή να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση για πολλές ερωτήσεις. Κύριε Βανίστερόι, να σας καλησπερίσω καταρχήν, σας ευχαριστώ. Μιλήσατε για την πολιτική, αυτή την επικοινωνιακή. Υπάρχει μία ε, θετική εξέλιξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μιλήσατε επίσης και για μία εταιρικότητα που υπάρχει στα πλαίσια της συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κινείται ως διευθυντήριο. Εμείς ε, κινούμαστε με βάση το επενδυτικό πρόγραμμα για την Ευρώπη. Μιλάμε για υψηλά αριθμητικά στοιχεία που δεν λένε τίποτα στους ανθρώπους καθεαυτά. αυτά. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κινηθούμε πέρα από το επενδυτικό πρόγραμμα σε μια πολιτική επικοινωνία σε σχέση με μεμονωμένα προγράμματα όπου βρίσκουν τη σωστή ανταπόκριση οι πολίτες. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Ο κόσμος έχει αλλάξει, Δεν έχουμε ούριο άνεμο πλέον. Έχουμε με τοπικούς ανέμους και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι πολίτες δεν είναι πάντα στο πλευρό μας πλέον. Και εδώ έχουμε να μάθουμε πολλά σε σχέση με το περιεχόμενο της επικοινωνιακής μας πολιτικής. Αλλά θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι χρειάζεται μία ευρύτατη συμμαχία, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από μόνη της δεν μπορεί να έχει το σωστό αντίκτυπο στην ε, κοινή γνώμη της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε μία διευρυμένη ε, συμμαχία και βεβαίως να κινηθούμε από κοινού Μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό φέτος, διότι οι 27 που θα συνεχίσουν σε αυτή την ε, κοινή περιπέτεια την πορεία τους, ε, γνωρίζουν ότι πρέπει να είναι ενωμένε αυτές οι χώρες, πρέπει να έχουν μια κοινή επικοινωνιακή πολιτική και να πούν στους πολίτες γιατί θέλουν να προοδεύσουν από κοινού. Και πρέπει να πείσουν και τους πολίτες να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευελπιστώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα υπάρξει κάποια αναγνώριση των μεγάλων σφαλμάτων του παρελθόντος που έγιναν από κάθε μορφή εκπροσώπησης, από δημόσια πρόσωπα, που στην ουσία ε, διεμβόλησαν τις Βρυξέλλες. Ελπίζω να μην ξαναγίνει αυτό. Ελπίζω όλοι να πούμε από κοινού τι πρέπει να γίνει για το μέλλον, να έχουμε μία ενιαία φωνή. Σε σχέση με την πρόταση ως προς τις ε, φυσικές καταστροφές, με, εκπλήσει, με εκπλήσουν αυτά που ακούω. Δεν ε, πιστεύω να υποθέτεται ότι εγώ θα απομακρυνθώ από την πρόταση της Επιτροπής. Με εκπλήσουν οι επικρίσεις η αλληλεγγύη δεν αφορά μία χώρα. Είναι μία αρχική και ουσιώδης αξία που είναι η πεμπτουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι φυσικές ε, καταστροφές μπορούν να πλήξουν και άλλες χώρες, όχι μόνο την Ιταλία και δυστυχώς ε, κάποια μέρα θα πλήξουν και άλλες χώρες. Γιατί λοιπόν να μην απαντήσουμε κατά τον ίδιο αλληλέγγυο τρόπο όταν μεμονωμένα κράτη-μέλη, ακόμα και η Ολλανδία, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ε, συνθήκες, παρόμοιες συνθήκες μεγάλης πίεσης. Δεν Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να προβάλλει μία πολιτική που να αφορά αποκλειστικά την Ιταλία. Ως προς τον, ε, τον τύπο μέτρων που προτείναμε, έχω να πω τα εξής. Πιστεύω ότι η, η Ευρώπη αναφέρεται και σε σύμβολα και Όταν υπάρχουν δεινές συνθήκες, η Ευρώπη θα είναι δίπλα στους πολίτες αυτούς που πρέπει να ξανασταθούν στα πόδια τους και θα πρέπει να χρηματοδοτήσει μέχρι τελευταίου ευρώ τα συγκεκριμένα μέτρα που σχετίζονται με τις φυσικές αυτές καταστροφές. Αυτό το σύμβολο έχει μεγάλη δύναμη και εδώ έγκυται και η αξία αυτής της πρότασης. Φυσικά θα πρέπει να ελέγξει κανείς κατά πόσο ορισμένες ε, βασικές αρχές ε, της ε, πολιτικής συνοχής διατρέχουν κίνδυνο. Πρέπει να υπάρχει πάντα έλεγχος. Και δεν θα εκτεθούμε όταν τα μεμονωμένα προγράμματα δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν ε, μια κατάσταση. Όπως είπε και η κυρία Νταμάτο, η πρόταση αυτή είναι ε, μία συγκεκριμένη πρόταση που αφορά τα έργα ανοικοδόμησης και αποκατάστασης και αυτό αφορά και την εθνική κληρονομιά της χώρας. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει κατάχρηση σε αυτή την περίπτωση από τα κράτη-μέλη σε σχέση με αυτή την συγχρηματοδότηση που ενέρχεται στο 100%. Αλλά θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα ως προς τα επιμέρους στοιχεία του για να απαντήσουμε σε αντιρρήσεις και αμφιβολίες. Επίσης θα ήθελα να απαντήσω με κάθε προσοχή και στα άλλα ερωτήματα της κυρίας Μάτο. γιατί δεν είναι θέματα που σχετίζονται με τη δική μου προσωπική ευθύνη, αλλά ως προς τον αποκλεισμό της δημόσιας ε, συγχρηματοδότησης, της δημόσιας χρηματοδότησης που σχετίζεται με τις φυσικές καταστροφές και την ε, σχετική οδηγία, η Επιτροπή μέσω του Προέδρου της έχει εκφραστεί επί του θέματος. Και αναφερθήκαμε για επιμέρους δαπάνες, τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε μεμονωμένα. Και υποβάλλεται και μία δεύτερη ερώτηση, την οποία δεν θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής. Πέρα από τη δημόσια χρηματοδότηση. Όχι, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Εντάξει. Εντάξει. Κυρία Κρέλ. Αναφερθήκατε ιδιαίτερα στην οδηγία Omnibus, στο κανονιστικό αυτό πλαίσιο και αναφερθήκατε και σε ορισμένες προτάσεις που, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο και αποτελούν ουσιαστική αλλαγή της διαρθρωτικής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής, με συγχωρείτε. Νομίζω ότι αναφέρεστε ιδιαίτερα στο εξής. Στο ότι μεμονωμένα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν για τη μεταφορά πόρων και ε, στο εύση και σε άλλα μέσα, αν κατάλαβα καλά. Η πρόταση αυτή θα ήθελα να τονίσω ότι περιορίζεται στην μία δυνατότητα και αυτή η δυνατότητα αφορά το κράτος μέλος και μόνον αυτό. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν δεν βλέπω ποια ουσιώδης αλλαγή θα γινόταν στην πολιτική συνοχής, εκτός αν τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο μέσο για την κατανομή αυτού του κονδυλίου. Αλλά δεν ξέρω διαφορετικά, δεν βλέπω πώς η πολιτική συνοχή πλήτεται. Κύριε Βέρνερ. Αναφερθήκατε και εσείς στα ίδια θέματα. Και το μνημπού στις δυνατότητες, δηλαδή μεταφορών από το ΙΣΕΦ. Και πιο συγκεκριμένα ρωτήσατε τα επιτεύγματα, τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής πώς μπορούμε να το διασφαλίσουμε στο πλαίσιο του έτσε. Δεν θα τα εξασφαλίσουμε. Δεν θα μπορούσαμε να τα εξασφαλίσουμε και δεν θα ήθελα εγώ να τα εξασφαλίσουμε. Ιδάλλως υπονομεύουμε την πολιτική συνοχή. Δεν σας αποκρύπτω ότι δεν ενθουσιάστηκα όταν άκουσα κάποιους ε, από αυτούς που σχολιάζαν το έτσι οι οποίοι επεσήμαναν τις γεωγραφικές ανισορροπίες. Μα το έτσι δεν είναι πολιτική συνοχή. Και αν κοιτάξει κανείς την κατανομή του, των κονδυλίων του έτσι συνολικά, είναι ε, σε μεγάλο βαθμό πιστή η αντανάκλαση του μεγέθους του ΑΕΠ. Μπορεί να μην έχει λοιπόν χαρακτήρα καθαρά αναδιανεμητικό το έτσι, αλλά ούτε και οδηγεί σε οπισθοδρόμηση. Με ενισχύει αυτό, όχι δεν με ενισχύει, γιατί αυτό είναι ο στόχος της πολιτικής συνοχής, δεν είναι ο στόχος του έτσι. Για το έτσι, ε, τα σχόλια δυστυχώς εκτός μικροφώνου. Άστο. Εμείς δεν επιβάλλουμε σε κανένα να δώσει χρήματα για το έτσι. Δεν κάναμε καμία πρόταση μεταφορά κονδύλιων από την πολιτική συνοχή στο έτσι. Ας είμαστε σαφείς. Δυνατότητα υπάρχει, γιατί θα να τη μέλη. Εκείνα θα αποφασίσουν δηλαδή. Τι θέλουν. Και αυτή νομίζω είναι και η κύρια διαφορά. Δεν υπάρχει ανάγκη, υποχρέωση δηλαδή μεταφοράς κονδύλιων από την πολιτική συνοχή στο έτσι. Και για να επανέλθω στην ουσιώδη συζήτηση που μας περιμένει. Τι είδα και γιατί σα είπα ότι δεν ενθουσιάστηκα όταν άκουσα κάποιους να σχολιάζουν ότι το έτσι δεν πρέπει να ακολουθεί την πολιτική συνοχή, να συμπεριφέρεται πιο πολύ στην πολιτική συνοχή γιατί πρόκειται για δύο διαφορετικά εργαλεία. Δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ίδιες προϋποθέσεις, ούτε στην ίδια λογική. Το έτσι ε, θεσπίστηκε για να ε, καλυφθεί το κενό των επιδοτής των ε, επενδύσεων στην Ευρώπη. Μακροοικονομικό εργαλείο είναι, ενώρο Η πολιτική συνοχή δεν επιδιώκει τον ίδιο στόχο. Επιδιώκει στρατηγικό προγραμματισμό. Η πολιτική συνοχή αφορά την λήψη υπόψη των αναγκών της κάθε περιφέρειας στην Ευρώπη. Επομένως, δεν, μας, ε, δεν αφορά την πολιτική συνοχή σε ένα μεμονωμένο πρόγραμμα, έργο, κατασκευή, αντίθετα με το έτσι. Και αυτή είναι η θεμελιώδη τους διαφορά. Θεμελιώδης διαφορά που θα πρέπει να συνεχίσουμε να τονίζουμε και στους επόμενους μήνες. διότι η Ευρώπη, με απολύτω πεπισμένο, χρειάζεται πολιτική συνοχή. Και το έτσι δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πολιτική συνοχή, διότι το έτσι ε, προσανατολίζεται στην εκτέλεση έργων. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε η θεματική συγκέντρωση, ούτε ο στρατηγικός προγραμματισμός όπως είπα, ούτε τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει η, η στόχευση συγκεκριμένο, συγκεκριμένη περιφέρεια, έκταση, επικράτεια, που είναι ο στόχος της πολιτικής συνοχής. Για, την, για τις περιφέρειες με καθυστέρηση ανάπτυξης, κυρία Κρέλ, φαίνεται ότι δεν είμαι αρκετά σαφής. Ας μιλήσω λοιπόν πιο απερίφραστα για τη Σικελία. Η πρόθεσή μας δεν είναι να αμφισβητήσουμε την ανάγκη να εξακολουθεί να προσφέρεται υποστήριξη στη Σικελία. Η πρόθεσή μας είναι με κάθε εντιμότητα να επιχειρήσουμε να αντιληφθούμε τι ακόμη πρέπει να κάνουμε για να έχουμε περισσότερη επιτυχία εν γέννη σε περιοχές όπως η Σικελία. Πιστεύουμε ότι υφίστανται διαρθρωτικά εμπόδια στη Σικελία, εμπόδια στην ανάπτυξή της, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επομένως, βασική ιδέα είναι να προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε την πολιτική της συνοχής με νέες διαστάσεις που θα βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτά τα συγκεκριμένα και διαρθρωτικά εμπόδια για να περάσουμε σε μια πιο επιτυχή ε, σύγκληση των περιφερειών. Όπως ε, ισχύει εν γέννη για την νότια γιατί βέβαια αφορά ολόκληρη την Νότια Ιταλία, όχι συγκεκριμένα τη Σικελία. Και βεβαίω ο στόχο είναι να δώσουμε και την ε, απάν, αποκρούσουμε τα επιχειρήματα εκείνων που λένε ότι δεν κάνετε καλά τη δουλειά τη πολιτική συνοχή, γιατί μπορεί καλέ να είναι οι προθέσει, αλλά εδώ και 30 χρόνια σε ορισμένε περιοχές δεν έχετε ε, παραγάγει ορατά αποτελέσματα. Πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση σε αυτές τις επικρίσεις. έκθεση συνοχής. Σας είπα ότι στόχος μας θα είναι όντως να εισαγάγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για να έχουμε πλήρη εικόνα στη μελέτη των μελλοντικών μας προτάσεων εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες προσθέτω. Επομένως αυτή είναι η πρόθεσή μας, επίπεδο και Διευθυνσίας για τις Περιφέρειες, αλλά σήμερα δεν είμαι σε θέση να σας πω ότι σε αυτή την απόφαση θα καταλήξει η Επιτροπή συλλογικά. Αντιλαμβάνομαι τις ε, ανησυχίες σας για το χρονοδιάγραμμα, για το πρόγραμμα. Είναι πολύ περιπλοκές οι εποχές που διανύουμε. Και μπορώ να προβλέψω ότι η Επιτροπή θα χρειαστεί με πολύ μεγάλη προσοχή να σχεδιάσει το χρονισμό ή ασδήποτε πρωτοβουλίας θα προτείνει την επόμενη διετία λόγω ακριβώς αυτής της ανάγκης, της επιταγής, της διαφύλαξης, της ενότητας των 27. Πρέπει δηλαδή να είμαστε βέβαιοι, να έχουμε την εγγύηση ότι στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Λυπή Ένωση, η Ένωση των 27, θα διατηρήσει τη συνοχή της. Με τον κύριο Νομίζω ότι δεν θέσατε περισσότερες ερωτήσεις ε, από τους υπόλοιπους ομιλητές. Σχολίασα τα των φυσικών καταστροφών σχετικά με, τις, ε, με τα λεγόμενα decommitments, τις απαλλαγές από τις υποχρεώσεις. Τα μέσα είναι διαθέσιμα, αλλά το θέμα αυτό ε, για το 2013 είχε τεθεί και φέτος θα τεθεί ακόμα περισσότερο όταν αρχίσουμε να κλείνουμε κάποια προγράμματα. Σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να προκαταλάβει ε, σε ποιο ε, ποσοστό θα φτάσουν ε, αυτές οι επιστροφές. Ότι προωθηθεί στον τελικό δικαιούχο μέσω των ενδιαμέσων και μέσω των χρηματοοικονομικών μέσων μέχρι τον μήνα Μάρτιο του 2017. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι κάτι το αποδεκτό με τον κανονισμό συμβατό, με τον κανονισμό 2007-13. Τους επόμενους δύο μήνες λοιπόν Έχουμε κάποιες δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασης. Και τώρα σχετικά για την εσωτερική συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως δεν πολύ κατάλαβα εκεί τη συζήτηση την οποία είχατε με τον κύριο Σμέτσα. Κοιτάξτε, θα πρέπει να υπάρξει μια σύμβαση ανάμεσα στις επιμέρους γενικές διευθύνσεις για να βελτιωθεί η συνέργεια ανάμεσα σε αυτές και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν μιλάμε σαν παράδειγμα για την επιδίωξη της αριστείας, αυτό ήταν και το, η ουσία του μηνύματος του κ. Σμίτς, αλλά μπορώ να τον ρωτήσω να μου πει τι ακριβώς εννοούσε. Πάντως το θέμα ήταν η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες γενικές διευθύνσεις. Εντάξει, τώρα θα ξεκινήσω με το δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Ο κύριος Βαλκάφσελ, ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λεμέτρη για την παρουσία του εδώ σήμερα το απόγευμα. Αναφέρθηκε και στο θέμα των φυσικών καταστροφών ο Γενικός Διευθυντής και στην έννοια της αλληλεγγύης που θα μπορούσε να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις κοινωνικές και οικονομικές που μπορεί να δημιουργηθούν. Ξέρετε ότι υπάρχει για τα θέματα αυτά και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, το οποίο δημιουργήθηκε με βάση το άρθρο 2 ε, του κανονισμού του 2014. Όταν δημιουργούνται λοιπόν τέτοιου είδους καταστροφές, φυσικές καταστροφές και ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Αυτό Αλληλεγγύης. Ε, εφόσον ξεπερνά το 0,6% του ΑΕΠ ή το 1,5% του εσωτερικού ακαθάριστου προϊόντος της κάθε χώρας. Το θέμα λοιπόν εδώ τίθεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο σχετικά με την Ισπανία σε περιοχές όπως η Μούρθια και η Βαλένθια, σε επαρχίες όπως το Αλικάντε, αλλά και στην ίδια την περιφέρεια της Μούρθια, υπέφεραν πολύ σημαντικές φυσικές καταστροφές πρόσφατα μετά από καταιγίδε, πλημμύρες, ε, ε, θυελώδεις ανέμους. Ιδιαίτερα στη Μούρθια υπήρξε ένας πολύ υψηλός αριθμός ε, κατοικιών οι οποίες έπαθαν ζημίες, ξεπερνούν τις 5.000 εφήγησαν πάνω από 100.000 άνθρωποι και πάρα πολλά χιλιόμετρα ακτής καταστράφησαν από την καταιγίδα αυτή. Μιας και λοιπόν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο αυτό αλληλεγγύης ε, λόγω του μεγέθους του ελαχίστου όπως είπαμε, αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο μέσο έτσι ώστε αυτοί οι πολίτες οι οποίοι είναι χιλιάδες να μπορέσουν κατά κάποιο τρόπο να μετριώσουν τις αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της καταιγίδα. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και κύριε κύριε Φιντά, ευχαριστώ που είστε εδώ. Λουξεμβούργιος δεν χρειάζεται να ε, ενημερωθώ για την προσθέμενη αξία για το Λουξεμβούργο, αλλά ούτε και για το Βέλιο βέβαια, της Ευρώπης. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει η παραπομπή σε μια μελλοντική ανακοίνωση για τα ε, προβλήματα, ενδιάμεση ανακοίνωση. Τι είδου αξιολόγηση, τι είδου προβλήματα σκοπεύετε να συμπεριλάβετε και τι αποσκοπείτε με αυτή την ανακοίνωση. και αν ε, επιληθούν αυτά τα διασυνοριακά προβλήματα. Κράτη που έχουν κοινή με παραμεθόριο ή περιοχές αυτών στην παραμεθόριο δεν θα ενισχυθούν και άρα δεν θα ενισχυθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτών. Και δεύτερη ερώτηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και στην Επιτροπή αλλά και στη δουλειά σας και γενικότερα νομίζω πρέπει να εξηγούμε πάντα τι κάνουμε στη δουλειά μας. Εσείς, ως Γενικός Διευθυντής μιας ε, διεύθυνση, Γενικής Διεύθυνσης που ασχολείται με την περιφερειακή πολιτική, είστε επικεφαλή πολύ καλών έργων. Πρόκειται λοιπόν και μια, για ένα τομέα πολιτική που πρέπει να έχει πρωτοπορό ρόλο και ταυτόχρονα να τον κοινοποιεί, να έχει την κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική στην Ευρώπη. Έχετε λοιπόν ε, κάποιο master plan στη Γενική Διεύθυνση για τις Περιφέρειες για τη χρηματοδότηση των καλών έργων, για τη διαχείρισή τους, που να μπορεί και να προβάλλεται στο, στην κοινή γνώμη. Βεβαίω, διαρθρωτική πολιτική, περιφερειακή πολιτική είναι το μίσο που θα πρέπει να ε, μπούμε με επιθετικό, επιθετικά επιχειρήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα εδώ. σα συγχαίρω για την ε, θέση την οποία έχετε καταλάβει, η οποία βέβαια είναι μια πολύ δύσκολη θέση, αλλά και πολύ σημαντική για τα επόμενα χρόνια. Αναφερθήκατε στο θέμα της εφαρμογής και είπατε ότι το 2017 θα υπάρξουν οι πρώτοι καρποί. Να μην ξεχνά ότι έχουμε στον τέταρτο χρόνο της δημοσιονομικών προοπτικών και θα πρέπει να δώσουμε μεγάλο αγώνα σε επίπεδο προϋπολογισμού. Και εσείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνετε μεγάλη μάχη και για την πολιτική συνοχή λόγω ακριβώς της μείωσης των πιστώσεων πληρωμών τις οποίες ε, υποστήκαμε το 16 και θα υποστούμε για μία ακόμη φορά το 17. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιτυχία. Ελπίζω να πετύχετε και εφόσον θέλετε την υποστήριξή μας, φυσικά και θα την έχετε. Ένα άλλο θέμα αναφέρεται στην πρόταση Omnibus. σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους. Ξέρετε ότι και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου τα δοκιμάσαμε αυτά. Τώρα πλέον μετά από τις αλλαγές στον κανονισμό έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με υποχρεώσεις, αλλά τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να λένε ότι έχουν πολλά προβλήματα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις Πολλές φορές ε, ε, τα στοιχεία βασίζονται στο input και όχι στο output όπως θα έπρεπε. Ελπίζω λοιπόν το θέμα αυτό να καταφέρετε να το συζητήσετε με τους δημοσιονομικούς ελεγκτές και να βρείτε μια λύση. Ένα τρίτο σημείο αφορά το στρατηγικό ταμείο επενδύσεων. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι κάτι το οποίο δεν ανταγωνίζεται την πολιτική συνοχής. Αλλά έχουμε εδώ ένα πρόβλημα. Το ΕΦΣΥ κλέβει ορισμένα προγράμματα από την πολιτική συνοχή και εμείς έχουμε έλλειψη έτοιμων προγραμμάτων στην πολιτική συνοχή. Το pipeline είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πολιτική συνοχή και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα βρούμε μεγαλύτερες, περισσότερες μορφές συνεργασίας και να μην κλέβουμε ο ένας από τον άλλο. Το τέταρτο θέμα αφορά το μέλλον. Εσείς υπογραμμίσατε αρκετά σημεία στην προσπάθεια την οποία έχουμε όλοι να κάνουμε στο μέλλον. θα πρέπει να δούμε όχι μόνο πώς συνδέονται τα θέματα αυτά με τις οικονομικές πολιτικές αλλά και με τις υπόλοιπες πολιτικές και πώς θα μπορέσουμε την πολιτική της συνοχής να τη συνδυάσουμε με τις υπόλοιπες πολιτικές του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Αυτά που μας είπατε για την αλληλεγγύη δεν θα τα επαναλάβω, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω πλήρως. Και η τελευταία ερώτηση θα είναι από, από μένα. Μας ενημερώσατε κύριε Λεμέτρα για την ανακοίνωση που είναι υποπροετοιμασία γιατί είναι εκ των προτέρων ευαισιμότητα όπως επίσης και για το επίπεδο εφαρμογής και ε, σε ποιο βαθμό αυτό συνιστά πλέον μία απέτηση για τα κράτη-μέλη. Όλοι γνωρίζουμε ότι ορισμένα από τα κράτη-μέλη δεν δέχονται ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Πήραν την πληροφορία την οποία έπρεπε τον μήνα Μάρτιο. Θα περιμένουμε μάλλον την ανακοίνωση τον μήνα Μάρτιο. Τι θα γίνει μετά. Πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πλήρως τους επόμενους δύο μήνες ε, τις μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι το τι περιμένετε από εδώ και πέρα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε κάποιες από τις συστάσεις αυτές πριν το Μάρτιο ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποια διαφορετικά πλάνα δράσεις; Τι θα γίνει από το Μάρτιο και μετά σε σχέση με την εξάντε αιρεσιμότητα. Γι' αυτό σας παρακαλώ ε, μια σύντομη απάντηση από πλευρά σας. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους σας, θα είμαι σύντομος. Για τον κύριο Βαρκάτσελ, νομίζω ότι κάναμε αρκετά μέσω της τελευταίας τροποποίησης του Ταμείου ε, Αλληλεγγύης σχετικά με ε, τις γρήγορες καταβολές. Ε, αυξήσαμε τις πιθανές προκαταβολές. Αυτό είναι κάτι το οποίο κάνουμε και σε αυτή ακριβώς τη φάση με την Ιταλία. Αναφερόμενος τώρα στην ανησυχία την οποία εκφράσατε, ότι δηλαδή τα ανώτατα όρια ε, για να μπορέσει να στηριχθεί κανείς, ότι είναι σε υψηλό επίπεδο, υπάρχει και ένα περιφερειακό κριτήριο το οποίο επιτρέπει και περιφερειακές καταστροφές να λαμβάνονται υπόψη εφόσον σε περιφερειακή βάση οι ζημίες είναι υψηλές. Συνεπώς λοιπόν, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε. Φυσικά υπάρχουν και τα θέματα των ορίων. γιατί πράγματι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποζημιώνει για την παραμικρότερη τοπική μικρή κλίμακας φυσική καταστροφή. Αλλά παρόλα αυτά, εάν έχει υπάρξει μια σοβαρή ζημία, αν έχει υπάρξει μια σοβαρή βλάβη, τότε το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι αυτό το οποίο έχει τη δυνατότητα να παρέμβει. Άρημον. Μιλάμε για μια ανακοίνωση η οποία ε, θα ολοκληρωθεί ε, τον ε, Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω ποια ακριβώς θα είναι η κατάληξη αυτής της διαδικασίας, αλλά σε επίπεδο αν θέλετε φιλοσοφίας και σε επίπεδο των προπαρασκευαστικών αν θέλετε βημάτων, αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσω ακριβώς και των δημοσίων διαδουλεύσεων είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το τι ακριβώς συνιστά τις συγκεκριμένες δυσκολίες για τις διαμεθοριακές προσπάθειες τις οποίες έχουμε αναλάβει ε, και για τη μετακίνηση των πολιτών και για τις μικρομεσαίες που προσπαθούν να απολύσουν τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους 20 χιλιόμετρα μετά τα σύνορα κτλ. Συνεπώς λοιπόν αυτό το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω προς εσάς σήμερα είναι ότι ήμασταν δεκτικοί για κάθε ε, είδους μαρτυρία αν θέλετε. Συνεπώς τα ευρήματα θα πρέπει να είναι ε, νομίζω αρκετά ενδεικτικά, αλλά δεν μπορώ να σας πω σήμερα ποιες θα είναι οι προτάσεις μας σε σχέση με την δημόσια δράση που θα πρέπει να αναλυθεί για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων. Σε επίπεδο τώρα ανακοινώσεων από πλευρά μας έχουμε μια δυσκολία στη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο. Πολύ σωστά είπατε ότι εμείς για πάρα πολλά προγράμματα ε, είμαστε η πηγή των γνώσεων που είναι απαραίτητες για να προχωρήσουμε και είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να υπάρξει αμφίδρομη επικοινωνία. Δεν ξέρω με τις με 400-500 διαχειριστικές αρχές που υπάρχουν για την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και την επιλογή των επιμέρους προγραμμάτων. Συνεπώς λοιπόν έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν ακριβώς και την καλύτερη ευκαιρία επικοινωνίας με τους πολίτες. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε σαφώς την κατάσταση Μέλετιτς. Για τα θέματα της εφαρμογής δεν έχουμε να πούμε πολλά. Ε, αναφερθήκατε σε μια κατάσταση ΚΑΤΣ 22 χωρίς ε, προφανή διέξοδο όταν μιλήσατε ε, για τις επιλογές οι οποίες υπάρχουν. Η πλειοψηφία των κρατών του Συμβουλίου δεν δέχονται ότι τα απλοποιημένα, οι απλοποιημένες επιλογές κόστους μπορεί να είναι υποχρεωτικές. Ενώ αναγνωρίζουν, αναγνωρίζουν ότι τελικά θα ήταν μια πάρα πολύ σοβαρή απλοποίηση και τελικά φοβούνται τον τρόπο με τον οποίο οι δικοί τους δημοσιονομικοί ελεγκτές θα κρίνουν την μέθοδο αυτή. Και αυτή είναι η δυσκολία την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Είναι μια διαδικασία μαθητείας θα έλεγα. Δεν είχαμε απλοποιημένες ε, τέτοιες μορφές κόστους ε, στο παρελθόν. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς ε, μέσω της ενθάρρυνσης αύξησης των επιπέδων εμπιστοσύνης ανάμεσα στις τοπικές ελεγκτικές διαδικασίες και στις κοινοτικές διαδικασίες, να ξεπεράσουμε αυτό το δίλημα της κότας και του αυγού ή του αυγού και της κότας. Να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο. Και θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπατε και για το εύση. Το θέμα δεν είναι ο ανταγωνισμός. Και δεν είναι ο ανταγωνισμός το θέμα. Ε, δεν είναι η κλοπή των προγραμμάτων. Οι διαφορές συνίστανται στην χρηματοδότηση ε, σύμφωνα με το ΕΦΣΥ, γιατί από τη μία έχεις να κάνεις με ένα δάνειο, από την άλλη έχεις να κάνεις με μια επιδότηση. Ε, αυτό δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και είναι κάτι που επηρεάζει τις επιλογές. Το πρόβλημα του να υπάρχουν ακριβώς pipeline επιλογής ισχυρά είναι κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο στο ΕΦΣΥ, αλλά είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους και ιδιαίτερα και υπό το φως της επομένης δημοσιονομικής περίοδου, γιατί είναι ένα από τα προβλήματα της αργής εφαρμογής. Πέρυσι τα κράτη-μέλη μας είχαν πει ότι είχαν υποβάλει 300 ε, μεγάλου μεγέθους προγράμματα. Και τελικά ε, το μόνο το 20% ε, κατετέθησαν ολοκληρωμένη πρόταση. Και η Πολωνία από μόνη της ήταν τα 40. Αυτά όλα δείχνουν λοιπόν ότι υπάρχει μια έλλειψη οριμότητας όταν έχουμε να κάνουμε με μεγάλα προγράμματα κυρίως υποδομών, τα οποία χρειαζόμαστε αλλά τα οποία δεν είναι προετοιμασμένα όπως πραγματικά θα έπρεπε να είναι. Και τώρα για τις αιρεσιμότητες, τις εξάντε αιρεσιμότητες. Η ανακοίνωση την οποία θα κάνουμε αναφέρεται στο χρησιμότητα ε, της συνολικής αξιολόγησης. Δεν θα δακτυλοδεικτήσουμε εμείς συγκεκριμένες αιρεσιμότητες οι οποίες είναι ακόμα και σήμερα ανεκπλήρωτες. Η επίσημη προθεσμία ήταν η 31η Δεκεμβρίου του 2016. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να αναφέρουν στην ολοκλήρωση αυτών των ερεσιμοτήτων τον Ιούνιο. Στην ουσία λοιπόν έχει υπάρξει μια παράταση εξαμήνου, αυτό το εξάμηνο, αυτή την κρίζα ζώνη αν θέλετε, ε, θα προσπαθήσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αν δημιουργηθούν θέματα, ξέρετε τι λέγει ακριβώς ο κανονισμός. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λεμέτρο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα σας ε, καλούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Ρέτζη, γιατί αυτό είναι ο καλύτερος ε, τρόπος να είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. We continue. Συνεχίζουμε. Um, Συνεχίζουμε τώρα και θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω την υπόθεση Omnibus. Τη γνωρίζετε πολύ καλά και θα ήθελα απλώς να αναφέρω ότι προετοιμάζουμε μία γνωμοδότηση δυνάμει του άρθρου 54 συν συν συν με, τις, ε, με βάση τις συγκεκριμένε αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι η επικεφαλής, ε, η επί της ουσίας η υπεύθυνη Επιτροπή Γι' αυτό κυρία Κρέλ είχε προετοιμάσει το πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων μέσα σε δύο-τρεις εβδομάδες. Ελπίζουμε να υποβάλει το προσχέδιο γνωμοδότησης τον επόμενο μήνα και να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Απρίλιο για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα του Κοινοβουλίου. Για να μην χάνουμε χρόνο, θα δώσω το λόγο στην κυρία Κρέλ για να μας πει για τις εξελίξεις του θέματος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όντως, ήταν με μετεμποδίων η εκκίνηση, ιδιαίτερα στο Κοινοβουλίο της, ε, του κανονισμού Omnibus. Θέλαμε εμείς από την Επιτροπή Περιφερειών τη δυνατότητα δύο γνωμοδοτήσεων. Μίας καταρχάς που θα αφορούσε καθαρά τον ε, κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής, το ΕΤΣΕ κτλ. και άλλη μία για τους δημοσιονομικούς κανόνες και οτιδήποτε άλλο βγαίνει έξω από την πολιτική συνοχής. Μάλιστα ήμασταν και σε συμφωνία με τους δύο συνεισηγητές, τον κύριο Αρτουή και την κυρία Γκρέσλε αλλά η διάσκεψη των Πρόεδρων άλλα αποφάσεις. δεν ξέρω γιατί ακριβώς, και μάλιστα μόλις πριν τα Χριστούγεννα, 15 Δεκεμβρίου, αν δεν απατώμε. Άρα χρειάστηκε σε μια έκτακτη ε, συνάντηση των συντονιστών να λάβουμε αποφάσεις για τα περαιτέρω. Και γι' αυτό έχω αναλάβει τώρα εγώ ως εισηγήτρια προσπαθώντας βεβαίως να ε, προετοιμαστώ όσο το δυνατόν πιο εντατικά για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για σήμερα. Εν πάση ειλικρίνεια θα σας πω ότι για ορισμένα σημεία δεν έχω ακόμη κατασταλάξει σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η γνωμοδότηση. Γι' αυτό θα χρειαστώ τη δική σας ε, υποστήριξη και τις ενδείξεις. Είναι πάντως διφλονοκούμενο ε, μη διαφιλονικού μονοτελείως το ότι θέλουμε απλούστευση του εις λειτουργίας του δημοσιονομικού κανονισμού. Πάντα αυτό ζητούσαμε ως κοινοβούλιο. Και δεν νομίζω να έχει κανείς αντίρρηση. Καμιά φορά διαβάζοντας την πρόταση της Επιτροπής, δεν μπορώ να πω ότι πείθομαι ότι απλουστεύει με τις προτάσεις της το κανονισμό. αλλά θα έχουμε και την ευκαιρία να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα, να λάβουμε εξηγήσει. Δεν έχω και εμπειρία από τράπεζα για να πω ότι ξέρω πώς χρησιμοποιούνται τα χρηματοοικονομικά μέσα. Θα χρειαστούμε και κάποιες συμβουλές από ειδικού. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα που μεταλανίζει. Ανέφερα εξάλλου μόλις ότι έχουν παρισπρίσει στοιχεία στη διαδικασία Omnibus που ξεπερνούν το στόχο της απλούστευσης και σε αυτά θα ήθελα να σταθώ λίγο. Στο δημοσιονομικό κανονισμό λοιπόν. Άλλωστε ανέφερε και νωρίτερα ο Γενικός Διευθυντής. Προτάσεις από την ομάδα εργασίας ψηλού επίπεδου Τώρα, βέβαια, μπορούμε να κάνουμε μόνο για την περαιτέρω δημοσιονομική περίοδο προτάσεις και πρέπει να προετοιμαστούμε για την προσεχή δημοσιονομική περίοδο να έχουμε έτοιμες προτάσεις για απλούστευση. Ιδιαίτερα λοιπόν, και ξεκινώ με αυτό, ε, ικανοποιεί το ζήτημα των απλούστευμένων δαπανών. υποχρεωτικά για τα έργα που δεν ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ ισχύει αυτός ο κανόνας, πολύ λογικός και θετικός. Βέβαια από διάφορες περιοχές, περιφέρειες, ε, ακούω ότι ακριβώς για τη νέα προγραμματική περίοδο έχουν ε, στριμωχτεί για να τηρήσουν με δύσκολους και περίπλοκους κανόνες ό,τι απαιτούσαν οι προηγούμενες διατάξεις και τώρα ξαφνικά είναι υποχρεωτική απλούστευση. Άρα θα χρειαστούν και άλλη δουλειά για την προετοιμασία. Το ξέρει πολύ καλά αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δεν περνάει από μια μέρα στην άλλη το σύστημα. Πρώτον λοιπόν γραφειοκρατική επιβάρυνση μεγάλη και μετά έρχεται η απλούστευση. Μήπως λοιπόν θα ήταν σκόπιμο να κοιτάξουμε να δώσουμε μια μεταβατική περίοδο. Ή να το προβλέψουμε σε βάση εκούσια. Όχι ε, υποχρεωτική σε μια πρώτη φάση. Θα πρέπει να μελετήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή είναι η ποια είναι η καταλληλότερη προσέγγιση. Όταν ξεκινάει μια νέα προγραμματική περίοδος, μερικές φορές παρουσιάζονται επιβραδύνσεις στη διατύπωση προτάσεων. Ε, ας μην οφείλεται σε αυτό. Να μην, επιβάλλουμε, να μην επιφέρουμε περαιτέρω καθυστερήσεις. Κατά αποκοπήν ποσά. Αυτά θα πρέπει όντως να αφορούν κάθε κράτος μέλος χωριστά με τις συγκεκριμένε προϋποθέσεις που το αφορούν και ξέρω ότι δεν μπορούμε να υποτιμούμε τις ε, ε, προσπάθειες και των εθνικών αρχών για να τηρήσουν τους στόχους της συνοχής. Δεν μπορούμε να τους βάσουμε παραπάνω προσκόμματα. Μέχρι στιγμής πάντως καλά. Δημοσιονομικά μέσα. Απλούστευση. Κρίθηκε απαραίτητη. Εισήχθη. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει ιδιαίτερως να μας απασχολήσει το πώς μπορούμε να αξιοποιούμε τα δημοσιονομικά μέσα. Με χαρά διαπιστώνω ότι η Επιτροπή έχει κάνει τις σωστές προτάσεις, γιατί άλλωστε και για την ίδια θα είναι χρήσιμα τέτοια δημοσιονομικά ε, μέσα σε σχέση με τα κρατημέλη. Αλλά όπως είπα, κάποιες ευκρινήσεις θα χρειαστούν. Το δεύτερο και από εδώ θα αρχίσω ουσιαστικά. Αλλαγέ στην πολιτική συνοχή, εκ των οποίων η πρώτη, την οποία και απεριόριστα υποστηρίζω, αφορά την πρόταση για μια νέα προτεραιότητα. Μέτρα για τους μετανάστες και του άσυλο. απλουστευμένη διαδικασία εταιρική σχέση, ε, τροποποίηση λειτουργικών προγραμμάτων, όλα αυτά προσδερούσε στο γενικό κανονισμό, πολύ σωστά, πολύ καλά. Ευέλικτη λοιπόν δυνατότητα αντίδρασης στις ανάγκες αυτές και για μένα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεύτερη πρόταση. Το είδαμε και στην προηγούμενη συζήτηση διασύνδεση της πολιτικής συνοχής με το, ε, ε, με το σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων του Juncker, το έτσι. Και εδώ έχω μεγάλα, μεγάλα ερωτηματικά. Και δει. Είχε πολύ μεγάλο συμβολισμό βεβαίως ο σχεδιασμός του σχεδίου Juncker και για κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, αλλά πάνω απ' όλα για εγγυήσει χάρη στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό που θα αποδέσμευαν κονδύλια, δημόσια κονδύλια για μεγάλα έργα που θα προχωρούσαν σε συνεργασία των μελών και επιτροπής έργων που δεν θα μπορούσαν τουλάχιστον δεσμευτικά να προκύψουν χάρη στην πολιτική της συνοχής με προσέλκυση ταυτόχρονα και ιδιωτικών επενδύσεων εκεί όπου τα κονδύλια, εφόσον τα κονδύλια από τον, ε, τους δημόσιους προϋπολογισμούς δεν αρκούν ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Ακροδών Μελών. Και τώρα τι κάνουμε στην πρόταση αυτή για τη διαδικασία ομνίμπους της Επιτροπής. πάλι βάζουμε το χέρι στο δημόσιο ταμείο, χρησιμοποιούμε δηλαδή κονδύλια του Δημοσίου Προϋπολογισμού, ένα κεντρικό εργαλείο για τα κράτη-μέλη και προσφέρουμε και πάλι εγγύησει. Γιατί πρέπει η ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεύτερη εγγύηση για τέτοια έργα. Πρώτο ερωτηματικό και πολύ σημαντικό. Γιατί να χρειάζεται κάτι τέτοιο. Τώρα δεν πρόκειται να επισέλθω σε συζήτηση για το τι εναλλακτική θα είχα να προτείνω, αλλά πάντως σε αυτό πρέπει να διατυπώσω ε, απορία και αμφιβολία. Δεύτερον, βεβαίως θα πρέπει να εγγραφούνται τα κονδύλια αυτά σε ένα κεντρικό εργαλείο, ε, νομοθέτημα, που, ε, στο οποίο θα προσφεύγουν τα κράτη-μέλη. Η εκτέλεση θα γίνεται βέβαια με την ε, συμμετοχή όλων μας και την υποστήριξη. Θα μπορούν όμως οι πάντες να έχουν την ίδια πρόσβαση, την ισότιμη πρόσβαση για όλους. Και εδώ ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Γιατί κανονικά τα κράτη-μέλη τα μέσα της συνοχής θέλουν να τα χρησιμοποιούν για τη συνοχή, για τους στόχους της συνοχής. Για μένα είναι απολύτως ασαφές το πώς θα διευθετηθεί αυτή η διαδικασία. Οι περιφέρειες, οι τοπικοί εταίροι θα συμφωνήσουν. Γιατί θα προπτεί για κονδύλια που θα βγαίνουν από τον κοινό κορβανά. Και σε περίπτωση εμφιβολίας θα συμφωνήσουν τα κράτη να πρέπει να περάσουν από την έγκριση επιτροπής για 500 εκατομμύρια φερρυπίν που θα χρειάζονται να περάσουν από ένα land της Γερμανίας για ένα έργο που αφορά μια περιφέρεια για να εκτελεστεί. Έτσι για μένα εδώ το ζητούμενο δεν είναι απλώς η άντληση κονδύλιων από την ε, πολιτική της συνοχής αλλά η εξασφάλιση δομών που αγωνιστήκαμε να εξασφαλίσουμε στην πολιτική συνοχή για πολλά χρόνια. Η εταιρική αρχή δεν έπεσε ως μάνα εξ ουρανού. Αυτές οι αρχές τώρα βλέπουμε να υπονομεύονται, εν πάση περιπτώσει να χαλαρώνουν οι προποθέσει τους. Χωρίς να είμαι και βεβαία ότι θα ικανοποιήσουν τον άλλο στόχο. Πάντως σίγουρα δεν θα είναι ε, εκείνοι που τα διαχειρίζονται τόσο ευαίσθητοι στα θέματα της συνοχής. Γιατί αν ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν ε, ε, μερικά εκατομμύρια, μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια από τον προπολογισμό της, της συνοχής για ένα άλλο έργο και μετά καλά εντάξει λίγο αργότερα θα τα φέρουμε πίσω χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της συνοχής, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Και οπωσδήποτε δεν μπορεί να είναι αυτό η πρόθεσή μας. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να αυτή η πρόθεσή μας. Με ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερος τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι, τι συμβουλές έχουν να μου δώσουν για, την περαιτέρω, για τις περαιτέρω επιλογές στην έκθεση. Πότε λοιπόν, ποιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων για να έχουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΣΕ. Πάντως σίγουρα όχι με την πρόταση όπως την έχει καταθέσει η Επιτροπή. Επίσης, τον τελευταίο κοινό κανονισμό που έχουμε παρακολουθήσει μαζί με τον ε, Λάμπρεχτ Φανίστηλ Ροή, τουλάχιστον σε 100 συνεδριάσεις συνδιαλλαγής με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, έχουμε νομίζω συμφωνήσει σε αυτό ότι υπάρχουν σημεία της διαδικασία Omnibus για τα κοινά προγράμματα δράσης, ότι ναι, θα ήταν καλό να αξιοποιούνται νέες καινοτόμε ιδέες, καλές ιδέες πρέπει να υποστηρίζονται. Αλλά αυτή η αρχή δεν εφαρμόζεται, δεν υλοποιείται στα κράτη-μέλη κατά πάσα πιθανότητα γιατί τους φαίνεται πολύ περίπλοκη. Και έτσι εδώ έρχεται η Επιτροπή αντιδρώντας να κάνει κάποιες προτάσεις, αλλά πάλι επισημένω στους συναδέλφους της Επιτροπής ότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με απάλληψη ορισμένων από τις αρχές που ήταν πολύτιμες για μας, την Επιτροπή μας ιδιαίτερα αλλά και όλο το Κοινοβούλιο. Φερρυπίν στο άρθρο 106 ζητήματα ε, ισότητας ευκαιριών, ευκαιριών και διακρίσεων. Φεύγει αυτό. Στον ε, κατάλογο επιλεξιμότητας Μπορεί αυτό να φαίνεται ότι διευκολύνει τις αποφάσεις γιατί τις καθιστά πιο απλές. Αλλά η πολιτική στόχη που έχει υποστηρίξει το Κοινοβούλιο, τουλάχιστον σε αυτό θέλουμε κάποιες διευκρινήσεις. Και παίρνω στο πρώτο τελευταίο σημείο που με ταλανίζει, γιατί εξίσου ε, σημαντική είχαμε ε, θεωρήσει και την υποστήριξη έργων στον χώρο του πολιτισμού, υποδομές πολιτισμού και τουρισμού. και ήρθε η ώρα στερα από μακρές συνομιλίες να συμφωνήσουμε για υποδομές μικρής κλίμακος για τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Τι σημαίνει το μικρής κλίμακος, μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ, κατεξαίρεση μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ, ε, επίπεδα χρηματοδότησης που μας φάνηκαν επαρκή. Και τώρα μαθαίνω ότι και από τα κράτη-μέλη αλλά και από κάποιους βουλευτές εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, διατυπώνεται έντονα το αίτημα να καταργηθεί αυτό ο φραγμός των 5 ή 10 εκατομμυρίων. Και θα σας πω ότι εδώ προβληματίζομαι σοβαρά. Γιατί ήταν ε, σοβαροί οι λόγοι για τους οποίους είχαμε πιέσει να αλλάξει η πολιτική της συνοχής ε, για να υποστηρίξει την καινοτομία, την ανάπτυξη τεχνολογίας, την έρευνα. Θέλαμε μια πολιτική συνοχής σύγχρονη. Και έχει εντωμεταξύ μειωθεί ο προπολογισμό, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί το ΆΠΑΝ στην προσεχή ε, προγραμματική περίοδο και θα το πω και κάπως προκλητικά, δεν θέλουμε να δώσουμε χρήμα στις ε, αρχές πέτρες, αλλά στα νέα μυαλά. Έτσι είχαμε πει τουλάχιστον. Το ερώτημα είναι παραμένει αυτή η επιλογή. Βεβαίω και καταλαβαίνω και μάλιστα να το δούμε και σε συνδυασμό με, την, ε, με το καταστροφικό σεισμό στην Ιταλία. Βεβαίω και υπάρχει ανάγκη να προσφέρουμε υποστήριξη. Αλλά διαρωτώ με το να καταργηθεί κάθε όριο πράγματι βοηθάει. Δεν θα πρέπει να ορίσουμε ένα το όριο που θα ήταν απαραίτητο και ενδεχομένως ένα μέσον διευκόλυνση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κράτους μέλους και Ευρωπαϊκής Επιτροπής των υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες να ξεπερνάει το όριο αυτό η χρηματοδότηση. Δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοι άρχισαν να με μισούν ήδη αλλά κάποια συμβουλή θα μου δώσετε κι εσείς. Άλλο ένα σημείο. Και θα παρακαλώ την Επιτροπή να το επαληθεύσει. Και μάλιστα για σήμερα περιορίζομαι μόνο όσον αφορά τα θέματα της δικής μας Επιτροπής. Ωστόσο στην τροποποίηση των δημοσιονομικών κανόνων βλέπω ένα σημείο το οποίο έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για μένα γιατί πάντοτε λέγαμε ότι θα πρέπει να οργανωθεί έκτακτο η ρύθμιση που θα καλύπτει μη επιστρεφόμενο φόρο προσθέμενης αξίας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής στα ε, έργα τα οποία υποστηρίζουμε. Και τώρα βλέπω στο άρθρο 180-4 μια διατύπωση που δεν φαίνεται τόσο ξεκάθαρη. Η εξαίρεση αυτή που προβλέπεται να συνεχιστεί στον χώρο της συνοχής. Αν μπορούν οι συνάδελφοι που καταλαβαίνουν καλύτερα αυτά τα οικονομικά θέματα από μένα να τα επαληθεύσουν, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πιστεύω. Κλείνοντα, θα σα πω ότι θέλω όσο δυνατόν πιο γρήγορα να επεξεργαστώ τι προτάσει αποτελεσματικά, ασφαλώ, χωρί όμω καμία χρονοτριβή. Ε, ωστόσο, δεν μπορώ να δώσω και καμία υπόσχεση. Πρόκειται για μια προσέγγιση πολύ σοβαρή της κυρίας Γκρέσλε ιδιαιτέρως τα θέματα αυτά, θέματα περίπλοκα και σε τόσο περίπλοκα θέματα πρέπει να αφήσουμε το χρόνο, το χρόνο του, να συζητήσουμε όλα τα σημεία και βεβαίως θα έχουμε και πυκνό χρονοδιάγραμμα ασφαλώς για να προλάβουμε χωρίς όμως να είμαι βεβαία ότι θα καταφέρουμε να ε, καταλήξουμε σε μια κοινή γραμμή η οποία θα είναι και εύκολο να υποστηριχθεί από τα κράτη-μέλη στον τριμερή διάλογο. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά ήδη για την όποια συνεργασία είχαμε μέχρι τώρα και βέβαια προσβλέπω σε περαιτέρω αποτελεσματική και επικοδομητική δημιουργική συνεργασία με τους ηγητές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. ε, συμμεριστείτε τα προβλήματα και τις αμφιβολίες σας ε, μαζί μας και θα ήθελα τώρα οι σκιώδεις να μας πούνε τι σκέφτονται. Ίσως έτσι θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα γίνει καλύτερο ή χειρότερο αυτό το πλαίσιο. Ε, ε εφόσον είναι κάτι το δύσκολο πρέπει να βελτιωθεί γιατί πρόκειται για ε, κάτι το περίπλοκο και τονίσατε ορισμένα προβλήματα που υφίστανται και σημεία που έχουν μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να δούμε όχι μόνο το περιεχόμενο, αλλά και τη θέση της Επιτροπής μας, γιατί μιλάμε για αποκλειστική αρμοδιότητα να μπορέσουμε να πούμε εμείς ναι ή όχι για θέματα που μας βρίσκουν σύμφωνους ή όχι. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει από τα πρώιμα στάδια να δούμε ποιες είναι και πού είναι οι κόκκινες γραμμές μας. Γιατί το ζήτημα αυτό μπορεί πράγματι να συζητηθεί εκτενώς. Αλλά ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε πριν πάμε στην ε, Ολομέλεια, κατά πόσο θα μπορέσουμε να έχουμε ε, διαλευκάνει κάπως τα πράγματα. Να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει μία προσέγγιση, μία σωστή προσέγγιση και μία προσέγγιση ως προς το Omnibus σε αυτή τη φάση. Θα πρέπει να μας πείτε δηλαδή εσείς ποια είναι τα σημεία στα οποία δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε στην προσέγγισή μας. Ως προς τα υπόλοιπα, νομίζω ότι κάνατε μία βαθύ κατατατή ανάλυση και νομίζω ότι έχουμε την ίδια προσέγγιση και εμείς. Ε, όταν μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας θα δούμε που βρίσκονται και οι δικές μας κόκκινες γραμμές. Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, όπως ξέρετε, πριν από 30 χρόνια ε, ήταν εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο λειτουργίας ως προς τους ε, χρηματοοικονομικούς κανονισμούς. Γιατί εδώ έχουμε κοινέ διατάξεις για τα διαφορετικά ταμεία και κοινού κανονισμούς για την εξωτερική μας δράση. Επειδή το χρηματοοικονομικό πακέτο είναι περίπλοκο, έχει επιβραδυνθεί η διαδικασία απόδοσης διαρθρωτικών πόρων. Γι' αυτό και υποστήριξα αυτή την αναθεώρηση κανόνων. Μέσα σε 15 ξεχωριστά έγγραφα για τα μακροχρόνια προγράμματα. Οι κανονισμοί που αφορούν τομεί έχουν νόημα έτσι ώστε η λήψη αποφάσεων να επιταχυνθεί. Γι' αυτό συνεχίσαμε να καταβάλουμε προσπάθειες για να μην υπάρχουν πια στενοποί και να φτάσουμε σε συνέργειες μεταξύ ΕΦΣΙ και άλλων διαρθρωτικών ταμείων, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος και οι δαπάνες, καθώς και ο αριθμός σφαλμάτων. Έτσι θα έχουμε ένα πιο ευέλικτο σύστημα δημοσιονομικών κανόνων που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει τάχιστα σε απροσδόκητες καταστάσεις ως προς τους δικαιούχους, νομίζω ότι από το απλουστευμένο αυτό πλαίσιο θα μπορέσουν να ευεργετηθούν. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα και Ε, έτσι οι δικαιούχοι θα εστιάσουν την προσοχή τους ε, στην ουσία των ζητημάτων για να μην υπάρξουν και περαιτέρω σφάλματα καθώς και παρατυπίες. Έτσι οι δικαιούχοι θα μπορέσουν να φτάσουν σε συμφωνίες και θα απλουστευτεί η διαδικασία και ως προς το διοικητικό άχθος και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Σε μια τέτοια περίοδο κρίσης θα πρέπει οι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες έτσι ώστε τα διοικητικά όργανα, οι υπηρεσίες να συμμετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Οι πολίτες θα πρέπει να νιώσουν ότι συμμετέχουν στο γίγνεσθε ε, της ευρωπαϊκής διαδικασίας. Θα προσπαθήσω κι εγώ με τη σειρά μου να σας πω πώς βλέπω το όλο ζήτημα από πλευράς φιλελευθέρων. Καταρχήν δέχομαι την ανάλυση που μας υποβάλλατε και θα πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι ο κύριος Βανίστελ Ρόι έχει δίκιο θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής μας για να φτάσουμε σε μία γνωμοδότηση. Θέλαμε να προετοιμάσουμε δύο γνωμοδοτήσεις, αυτό δεν στάθηκε δυνατόν. Θα μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε για το συνολικό πλαίσιο της πρότασης Omnibus, αλλά από πλευράς ε, Ρέτζι δεν πρέπει να απαρνηθούμε τις αποκλειστικές μας αρμοδιότητες. Υπ' αυτή την έννοια, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η απλούστευση. Θα πρέπει να την υπερασπιστούμε παντού, ακόμα και στο δημοσιονομικό μέσο. Αυτό μας έχει απασχολήσει επί μακρόν. Και τώρα ήρθε η στιγμή όπου μπορούμε να συμπεριλάβουμε την ε, πραγματική απλούστευση όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι το 2020. Επίσης, όταν ε, μιλάμε για το ΕΦΣΥ, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει και πάλι να δούμε τι θέλουμε. Γιατί όλες οι συζητήσεις περί κοινής ε, εργασίας, περί συνεργασίας και συμπληρωματικού χαρακτήρα των διαρθρωτικών ταμείων και του ΕΦΣΥ και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά είναι συζητήσεις. Συζητήσεις που γίνονται εδώ και αλλού. Αλλά τώρα ήρθε η στιγμή που θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι θέλουμε από αυτά τα μέσα. Δηλαδή δεν πρόκειται για ε, μέρος της πολιτικής συνοχής, αλλά για ένα διαφορετικό μέσο που αφορά τις περιφέρειες, το ευρωπαϊκό έδαφος. Υπάρχει συμπληρωματικός χαρακτήρας, αλλά και διαφοροποίηση του ΕΦΣΥ και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι το ε, χαρτοφυλάκιο αυτό, το Omnibus, δεν αφορά μόνο την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά προετοιμάζει και το μελλοντικό και η θέση της Ρέτζη θα πρέπει να αποτελέσει βάση εργασίας για το επόμενο πολιετές. Γι' αυτό ως κοιόδης πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις αρμοδιότητες της Ρέτζη, να μιλήσουμε για διαδικασία απλούστευσης, γιατί αυτό είναι το βασικό μήνυμα και να είμαστε πολύ σαφείς σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τα άλλα δημοσιονομικά μέσα ως προσαλλαγές ε, για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Βεβαίως είναι αλλαγές ε, όπου θα πρέπει να δούμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Θα δεχτούμε και τα μηνύματα του Συμβουλίου αλλά η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να δούμε ποια μέθοδο θα ακολουθήσουμε για να συμπεριλάβουμε τους κανόνες αυτούς στο λειτουργικό μας πρόγραμμα. Και φυσικά τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν για τα παρελκόμενα. Αυτά είναι τα πρωταρχικά μου σχόλια, αλλά νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ομερουσέ ε, δεν είναι εδώ, κυρία Βάνα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και κυρία Συγκητρία. νομίζω ότι ξεκάθαρα μίλησα για την επικριτική και απορριπτική ουσιαστικά στάση των πρασινών απέναντι στην προσέγγιση ομονιμπού τη Επιτροπής. Θα ακολουθήσουμε τι στάσεις σε μεγάλο βαθμό. Το θέμα για μας δεν είναι μόνο η προσέγγιση, ότι δηλαδή θα πρέπει εξάπαντο οι εμπλεκόμενες επιτροπές να μην ακροτηριάζονται, για να το πω και να μπορούν να συμμετέχουν στην επεξεργασία ενός ε, θέματος που δεν βλέπουμε εδώ να συσχεύει από πλευρά Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά και η δυνατότητα της ε, ανεπιφύλακτης και απεριόριστης μεταφοράς κοντιλίων για το έτσε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι αυτό θα σημάνει το τέλος της πολιτικής συνοχής. Γιατί βέβαια πάντα μας λένε και διαρριχνούν τα ηματιά τους ότι το έτσι δεν είναι ανταγωνιστικό της πολιτικής συνοχής, δεν την υποκαθιστά, πρόκειται για διαφορετικό εργαλείο. Αλλά δεν ισχύει αυτό 100%. Γιατί φαίνεται να προτιμά η Επιτροπή ρητά, τουλάχιστον αυτό το βλέπουμε στον κανονισμό Omnibus ε, πλέον, να διαγράφεται αυτή η προτίμηση της ε, Επιτροπής υπέρ του έτσι και κατά της συνοχής. Και αυτό το είδαμε και στις διευκρινήσεις που δοθήκανε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη για την ε, μεταφορά των πόρων από το η συνοχή προς το έτσε. Και επίσης η Συμβουλή των κρατών μελών στα έτσε θα αποκλείεται από τα κριτήρια του, ε, του υπολογισμού του κρατικού ελλείμματος. Δεν ισχύει αυτό και κανένα άλλο τομέα πολιτικής. Τι είδους λοιπόν ισότητα αντιμετώπισης μας λένε ή ότι δεν υπάρχει σαφής προτίμηση του έτσε για τις επενδύσεις ή ότι δεν αποτελεί το έτσε απειλή ή ότι δεν θα οδηγήσει αποδυνάμωση της πολιτικής της συνοχής. Δεν θα συμφωνήσω λοιπόν σε αυτό. Μια ερώτηση έχω ως προς την ουσία που δεν είδα να διευκρινίζεται, ως προς το περιεχόμενο περισσότερο, γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώ τι μπορεί να σημαίνει αυτή η πρόταση. Το shared implementation, ε, κοινή εφαρμογή αντί για κοινή διαχείριση, αντί για shared management. Να μας εξηγήσει η Επιτροπή παρακαλώ τι εννοεί και τι σημαίνει αυτό το shared implementation αντί για το shared management. Θα είναι διαφορετική η βάση, θα είναι διαφορετικοί η κανόνες, ενδεχομένως να μας δώσει και μερικά παραδείγματα πρακτικά. Βεβαίως και προσβλέπω με χαρά στην ε, συνεργασία και μέσα σας βεβαίως ε, κυρία Συγκήτρια, αλλά με όλες τις ομάδες, γιατί στη Ρέτζη έχουμε εδώ ε, από όλες τις ομάδες κοινή προσέγγιση και αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε τα όσα διεκδικήσαμε και με αγώνες εξασφαλίσαμε για τη συνοχή, για το, η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, ε, για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Όλες αυτές τις δεκαετίες αγώνων θα χαθούν. Και σε αυτό πιστεύω ότι ανεξαρτήτως κομματικών ε, χρωματισμών και αποχρώσεων θα σταθούμε όλοι απέναντι σε αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή, ή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διορθώνει ξανά ο προ, η πρόεδρος για τρίτη φορά, συγγνώμη, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Έχουμε ίσως καθυστερήσει λίγο. Και δεν νομίζω ότι μπορώ να καλύψω όλες τις πλευρές ε, του πακέτου Omnibus μέσα σε λίγα λεπτά. Να αναφερθώ όμως σε κάποια στοιχεία στα οποία ήδη αναφερθήκατε και τα οποία μπορεί να είναι ενδεικτικά για τον τρόπο σκέψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απλοποίηση, το είπε η κυρία Κρέλα, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε συγκεκριμένους στοχευμένους χώρους στο εσωτερικό του ESI, όπου θα μπορέσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα τώρα, στην περίοδο δηλαδή 14-20. Παράδειγμα, ο κανονισμός Ούμνιμπους δεν έχει σαν στόχο να απλουστεύσει την προγραμματική διαδικασία, διότι έχει ήδη εξελιχθεί. Οπότε δεν υπάρχει νόημα να το κάνουμε αυτό. Αυτό το οποίο όμως προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φτάσουμε σε μια ταχύτητα, αν θέλετε, κρουαζιέρας και επιδόσεων, την οποία ακόμα δεν έχουμε πετύχει θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε στο μέσο μιας προγραμματικής περίοδου χωρίς, και το επαναλαμβάνω αυτό, το υπογραμμίζω αυτό, χωρίς να υπονομεύσουμε τις διαδικασίες τις οποίες έχουν προβλέψει τα κράτη-μέλη. Δεν θέλουμε να ανατρέψουμε τίποτα στο μέσο της διαδικασίας. Γι' αυτό ακριβώς ε, οι περισσότερες ε, προτάσεις απλοποίησης στα πλαίσια του πακέτου Omnibus στην ουσία αυτό το οποίο κάνουν είναι να προσθέτουν επιλογές. Δίδουν νέες δυνατότητες χρήσης ελαφρώς τροποποιημένων ή και νέων μέσων προς όφελος της απλοποίησης, της απλούστευσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει ας πούμε τις προτάσεις μας. Σαν παράδειγμα, ε, τα, οι εναλλακτικέ επιλογές κόστους, οι καταποκοπήν πληρωμές ε, και για τα έμεσα κόστη και για τα άμεσα κόστη. Δίδουμε νέες επιλογές στο πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες και να μπορεί έτσι να καλύπτει τις μεμονωμένες ανάγκες κάθε προγράμματος. Υπάρχει μία εξαίρεση και αναφερθήκατε σε αυτό. Το απλοποιημένο κόστος θα είναι υποχρεωτικό για κάτω από τις 100.000. Αυτό ήταν μια άμεση αν θέλετε απάντηση σε ένα σημαντικό αριθμό παραπώνων εδώ και πολλά χρόνια για το υψηλό κόστος παράδοσης αν θέλετε των πιστώσεων αυτών διάθεσης των πιστώσεων αυτών και το ελεγκτικό κόστος ήταν ιδιαίτερα υψηλό, ιδιαίτερα για πολλά από τα μικροπρογράμματα τα οποία ξόδευαν περισσότερα χρήματα για τον έλεγχο παρά για το συγκεκριμένο, συγκεκριμένη επιδότηση. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να πάψει πλέον. Χρησιμοποιούμε το απλοποιημένο κόστος Ενθαρρύνουμε όλο και περισσότερα όργανα στα κράτη-μέλη να το κάνουν αυτό και για τα μικρά προγράμματα ας χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο αυτή αυτόματα, δημιουργώντας ένα πραγματικό streamlining. Τώρα, αυτά τα στοιχεία για τη μεταβατική περίοδο, η οποία τίνει να γίνει μόνιμη, Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια ε, ε, εναλλακτική μεταβατική περίοδος. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα πλέον. Να προσθέσω επίσης κάποια στοιχεία για τη σχέση ανάμεσα στο ταμείο, στα ταμεία μας και το ΕΦΣΥ, το Στρατηγικό Ταμείο. Νομίζω ότι σε επίπεδο ε, βασικό, γενικό καλύτερα, υπάρχει ανάγκη να είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία ανάμεσα στα δύο ταμεία, για τη σχέση ανάμεσα στα δύο ταμεία. Όταν σαν συνομοθέτες υιοθετήσατε τους κανονισμούς του ΕΦΣΙ, του ESI μάλλον, το ΕΦΣΙ δεν υπήρχε. Οπότε σε αυτή την περίοδο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα νέο σημαντικό επενδυτικό ταμείο το οποίο είναι εν λειτουργία και έχει άμεση σημασία θα έλεγα να δούμε ακριβώς πώς συνδυάζονται τα δύο ταμεία αυτά και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να τα συνδέσουμε καλύτερα και να χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις δύο πλευρές χρηματοδότησης. Συνεπώς θα ήταν λάθος αν δεν εξετάσουμε αυτή την δυνατότητα. Δεύτερον, ε, υπάρχει εδώ η σημασία της διασφάλισης της μέγιστης δυνατής συμπληρωματικότητας σε κάθε δημοσιονομική λειτουργία. Αυτό το έχουμε κάνει και σε άλλα ταμεία και για άλλα ταμεία και αυτό πρέπει να συμβεί και για το ΕΦΣΥ να υπογραμμίσω εδώ κάποια συμπληρωματικά στοιχεία μέσα από το ΕΦΣΙ και μέσα από το ESI. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σαν παράδειγμα, μπορεί να υποστηρίξει δραστηριότητες όχι από μόνη της, αλλά μέσα από το ESI ή μέσα από το Ταμείο ε, το Στρατηγικό. Αυτά θα επανέλθουν αργότερα σαν θέματα την ερώτηση της κυρίας Κρέλ για το ΦΠΑ θα το εξετάσουμε αυτό. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το άρθρο 180 αναφέρεται σε επιδοτήσεις άμεσου τύπου μόνον. Οπότε δεν τίθεται εδώ το θέμα της διαμοιρασμένης διαχείρισης ή της κοινής διαχείρισης. Τελειώνοντας να πω ότι εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε να βοηθήσουμε τη διαδικασία αποδοχής το ταχύτερο και το περισσότερο δυνατό. Όπως είπε και ο Γενικός Διευθυντής μου, υπάρχει ανάγκη έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν το πρόγραμμα αυτό να τεθεί σε λειτουργία και να έχουμε χρόνο ακριβώς να υποφεληθούμε και κατά τη διάρκεια της παρούσης, της μεσούσης προγραμματικής περίοδου. Συνεπώς λοιπόν ε, κάθε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας θα είναι χρήσιμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κρέλ να κλείσει τη συζήτηση. Ναι δεν μπορώ να πω ότι διαφωτίστηκα. Νομίζω ότι απέφυγαν οι πάντες με επιδεξιότητα τα πολιτικά ερωτηματικά που διατύπωσα, αλλά βέβαια έκαναν πάρα πολύ καλή ανάλυση. Εν θα προσπαθήσω να επεξεργαστώ μια καλή πρόταση. Ελπίζω να τα καταφέρω. Πριν έρθει η ώρα να κάνω την παρουσίαση στην Επιτροπή να συνομιλήσω και με τους κοιόδης. Πάντως βλέπω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για την απλούστευση στη γνωμοδότηση. Θα την υποστηρίξουμε από ό,τι βλέπω. Ίσως κάποια από τα περίπλοκα πολιτικά ζητήματα θα ήταν σκόπιμο να τα βγάλουμε από αυτή τη διαδικασία της γνωμοδότησης. Έτσι το λέω τώρα μου ήρθε ίσως μπορούμε να συνοηθούμε ότι κάνουμε μια, έναν διαχωρισμό ε, της θεματολογίας και βγάζουμε έξω από αυτή τη γνωμοδότηση το έτσι και τη συνοχή. Και περιμένουμε από την Επιτροπή να κάνει πιο συγκεκριμένε προτάσεις. Ίσως θα τις κερδίσουμε και χρόνο. ίσως έτσι να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε μια συμβαστική λύση. Έτσι μου ήρθε λοιπόν όπως σας είπα αυτή η ιδέα. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Ε, αυτά που σας είπα, πέραν του φόρου θεμένες αξίες ήταν του άρθρου 100, τι νούμερο 165, κάτι τέτοιο. Ε, αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. θα έχουν συνέπειες και στην απλούστευση εν γέννη του δημοσιονομικού κανονισμού, αυτή που θα προταθεί δηλαδή. Αλλά υπάρχουν θέματα που ανήκουν στις δικές μας αρμοδιότητες, θα πρέπει να απαντήσουμε. Ε, απλά ερωτήματα απλούστευση της πολιτικής συνοχής δεν θα είναι τα πιο δύσκολα θέματα για μας. Γιατί καιρό τώρα περιμέναμε πρόταση. Και τώρα πια θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Και εγώ θα προσπαθήσω να διατυπώσω στο δυνατόν πιο ουδέτερη και πρόταση το ταχύτερο δυνατό. Και σας ευχαριστώ θερμά. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτηση. Θα επανέλθουμε γρήγορα, τάχιστα. Θα σας υποστηρίξει και η γραμματεία όταν θα πρέπει να συνεδριάσουν ε, οι σκιώδεις. Δεν υπάρχει κάτι στα διάφορα. Η επόμενη συνάντηση, η συνεδρίες θα γίνει τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου από τις 3 το απόγευμα και μετά. Και τώρα κλείνει η ολομέλεια της ομάδας και θα ήθελα να αποχωρήσετε όλοι όσοι δεν είσαστε καλεσμένοι για τη συνάντηση των συντονιστών. Μόνο οι συντονιστές και ευχαριστεί και τους διερμηνείς η Πρόεδρος. Α, όχι, όχι, με συγχωρείτε, έχουμε διερμηνία μέχρι τις Άρα συνεχίζουμε με τους συντονιστές.